Κυρίε Κυρίες και κύριοι και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τώρα την επόμενη συνεδρίασή μας, το επόμενο πάνελ δηλαδή, για τη δημοσιονομική εξυγίανση βέλτιστες πρακτικές και το σύμφωνο, το δημοσιονομικό σύμφωνο. Έχω λοιπόν την ευχαρίστηση να σας απευθύνω το λόγο. Χαίρομαι πολύ που μπορέσατε να προσέλθετε στην συνεδρία αυτή την οποία οργανώνουν η Βουλή της Λετωνίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε να συζητήσουμε σημαντικά θέματα της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής διαχείρισης και των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Έχω σήμερα κοντά μου τους key speakers, τον κύριο Γιάννης Ρέις, Ρέιρς που είναι υπουργό Οικονομικών της Λετωνικής Δημοκρατίας. Έχουμε όμως και αντί του κυρίου Ντάισελ Μπλουμ, που είναι πρόεδρος της ε, Eurogroup ε, αυτός έχει άλλες ανηλυμένες υποχρώσεις ευτυχώς όμως έχουμε τον κύριο Ντόμινικ Χάνεγκαν που είναι μέλος της Ιρλανδικής Βουλής και πρόεδρος της ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδικής Βουλής. Έχουμε επίσης και τον Ευρωβουλευτή Όλη Ρεν, που είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω, ελπίζω ότι έρχεται, δεν είναι ακόμα εδώ. Στη σημερινή συνεδρία θα θα συμπροεδρεύσουμε αλλά πρώτα ένας μετά ο άλλος με τον ε, Ιταλό συνάδελφό μου κύριο Γκουαλτιέρη θα αρχίσω εγώ να κάνω και μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις ο ίδιος ο κύριος Γκουαλτιέρη θα αναλάβει τα ενία της συζητήσεως στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίας. Μερικές φορές είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε αυτές τις παραδοσιακές φράσεις των πολιτικών που δεν τις ακούμε καν όπως ε, λιτότητα, ε, μεταρρυθμίσεις, ανταγωνιστικότητα και δημοσιονομική εξυγίανση και ούτω καθεξής. Αλλά να με αφήσετε να σας θέσω υπόψη μια απλή σκέψη. Δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές αλλαγές είναι κάπως όπως σχεδιάζει κανείς και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για να μπορέσετε να περάσετε καλές διακοπές ή να έχετε καλή σύνταξη, έχετε λόγο να κόψετε κάποιες δαπάνες πριν. Να βρείτε μια καλύτερη δουλειά που να πληρώνετε καλύτερα δηλαδή και να, μην, και να αποφεύγετε να παίρνετε το καταλωτικά δάνεια και να κάνετε κάποιες αποταμιεύσεις για αργότερα μακροπρόθεσμα άλλωστε. Αυτό είναι το ίδιο και για τις ε, χώρες. Να εξετάζουν δηλαδή την αποδοτικότητα των δημοσίων οικονομικών και να προωθούν τους τομείς εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι δημοσιονομικές και άλλες διαθωτικές μεταρρυθμίσεις έδειξαν πόσο σκληρός είναι ο δρόμος αυτός, που όμως οδηγεί σε βιώσιμα αποτελέσματα. Αυτή πάντως η βιωσιμότητα είναι εύθραυστη. Σε ό,τι αφορά το αντιλήψη αποφάσεων, πιστεύω σε αποφάσεις που οδηγούν σε κάποια βιωσιμότητα. Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαθροτικές αλλαγές πρέπει να γίνονται όχι κατόνομα αλλά για να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα ε, του ε, ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου και ταυτόχρονα πρέπει να συνοδεύονται με καλά στοχευμένες πολιτικές που να επιτρέψουν την ανάπτυξη και την μείωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εκείνοι που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αυτά συζητούμε σήμερα και είμαι πεπισμένο ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ακόμα πολλά να διδαχτούν οι μεν από τις δε. Έχει νόημα να προσπαθήσει να μάθει κανείς κάτι από κάποιον που έχει ε, παρόμοιο τρόπο ζωής. Ελπίζω λοιπόν να είναι καρποφόρα η συζήτηση, να μας επιτρέψει να εξετάσουμε οι μεν τις ιδέες των δε όπως θα έπρεπε ίσως να κάνουν χώρες μέλη και στο μέλλον. Τώρα με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Όλι Ρεν που έφτασε. Ήδη έχω ανακοινώσει την παρουσία σας βέβαια πριν να έρθετε. Τώρα είμαστε πλήρεις εδώ και αν θέλετε μπορούμε να αρχίσουμε τις παρουσιάσεις των βασικών ομιλητών και με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Οικονομικών της Λετωνικής Δημοκρατίας, κύριο Γιάννης Ρεΐρς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρεν, κυρίες και κύριοι. Η Λετωνία έχει αναλάβει την προεδρία της, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη και δύσκολη περίοδο. Η Ένωση έχει πληγεί από χαμηλή ανάπτυξη και πολύ χαμηλό πληθωρισμό από πληθωρισμό σχεδόν. Και αυτά φαίνεται ότι θα συνεχίσουν ως τάσεις και στο μέλλον. Η ανεργία είναι ψηλή σε, έχει φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα. Η Κομισιόν και άλλες, άλλα διεθνή βήματα λένε ότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη στην Ένωση τα επόμενα χρόνια είναι πολύ χαμηλές. Η χαμηλή λοιπόν ανάπτυξη ισχύει από το 2008 τουλάχιστον και είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση γιατί όσο περισσότερο μένει η στασιμότητα τόσο πιο αναπότρεπτη γίνεται και μη αναστρέψιμη και χαμηλώνει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Οι αρνητικές, οι άσκημες οικονομικά αποτελέσματα θα θέσουν εν κινδύνο και το όραμά μας για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Παρά τα αρνητικά αυτά στοιχεία όμως, οι θεσμοί είναι διατεθειμένοι να βελτιώσουν τα πράγματα οικονομικά και επομένως ανέλαβαν ορισμένες σοβαρές πρωτοβουλίες και προτάσεις για να αποφευχθεί η στασιμότητα. Αν πιστεύουμε στην Ευρώπη ως πολιτική και οικονομική εντότητα παγκοσμίας, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και για να ανανεωθεί λοιπόν για να θερμανθεί οικονομικά η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική κυρίως δράση. Το σύμφωνο σταθερότητας και τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολλές απόψεις για το κατά πόσον οι πολιτικές λιτότητας είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των τρεχόντων αυτών οικονομικών προβλημάτων και για τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στη σταθερότητα των οικονομιών γενικότερα. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της κρίσης και ποιοι παράγοντες την εξηγούν. Πιστεύω ότι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εξηγούνται από πολλούς παράγοντες, συνδυασμό παραγόντων και από τις διαφορετικές οικονομικές δομές και κύκλους που αντιμετωπίζουμε, ιστορικούς λόγους και την εφαρμογή, τον τρόπο εφαρμογής ορισμένων δημοσιονομικών προγραμμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι με βάση όλους αυτούς τους παράγοντες και το γεγονός ότι υπάρχει ενιαίος χαρακτήρας της αγοράς μπορεί να υπάρχει και επίπτωση από το ένα κράτος στο άλλο. Άρα χρειάζεται μια συνδυασμένη λύση, ένας συντονισμός της οικονομικής πολιτικής για να μπορέσουμε να ταυτίσουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικονομικές ανισορροπίες και πού οφείλονται. Μια κοινή διευθέτηση δηλαδή που να αντιμετωπίζει τα βασικά στοιχεία όπως πρωτοβουλίες όπως πρόσθετες οικονομικές δαπάνες στους προϋπολογισμούς για λιγότερη και λιγότερη παράλληλα σπατάληση των πόρων. Αυτό σημαίνει μεταρρυθμίσεις και άρα αντιλαϊκά μέτρα ή μέτρα που δεν θα είναι δημοφιλή. Το σύμφωνο σταθερότητας θα μπορούσε να διευρυνθεί με τους εποπτικούς μηχανισμούς που είναι ουσιώδες στοιχείο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων έπειτα μείωση των ανισοτήτων μεταξύ χωρών μελών. Η Κομισιόν μπορεί να το αντιμετωπίσει αλλά κανένα άλλο όργανο δεν μπορεί. Μπορεί δηλαδή να γίνει μία ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών αλλά λίγα παραπάνω. Ξέρω ότι οι πολιτικές οικονομικές εξυγίανσης και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι κάτι πολύ δύσκολο και από πρακτικής και από πολιτικής και κοινωνικής απόψεως. Και αυτό το λέω διότι στη Λετωνία το ζήσαμε αυτό. Μπορεί μερικοί να έχουν αντιρρήσεις, αλλά η Λετωνία μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής περίπτωση, έτσι θα έλεγα. Το παρόν είναι πάντοτε αποτέλεσμα του παρελθόντος, αλλά το μέλλον εξαρτάται από τις τωρινές αποφάσεις που θα πάρουμε. Για τα δημοσιονομικά λοιπόν στις χώρες της Ένωσης πρέπει να δούμε τα εξής. Γενικά στους προϋπολογισμούς των χωρών μελών βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μια θετική τάση. Και για πρώτη φορά από το 2008 το έλλειμμα έχει κατεβεί στο κάτω από το 3% και αυτό νομίζω ότι θα ισχύσει και για τα επόμενα χρόνια στις περισσότερες χώρες. Επίσης θετικό είναι ότι η Κομισιόν ε, που είναι λιγότερο αισιόδοξη στις προβλέψεις της γενικά συμφωνεί με αυτά που δηλώνουν ή βλέπουν τα κράτη-μέλη. Για τα σχέδια προϋπολογισμού των χωρών μελών τα τελευταία αποτελέσματα της Κομισιόν είναι σαφή. Ουδέτερο το αποτέλεσμα για το 14 και το ίδιο προβλέπεται και για το 15. Αυτό βέβαια μπορεί να εξηγηθεί λογικά. Αλλά υπάρχουν και ανησυχητικά στοιχεία διότι πολλές χώρες μπορεί να μην φτάσουν στα επίπεδα που απαιτούνται για τη σταθερότητα όπως προβλέπει το σύμφωνο. Χαίρομαι γιατί σε με πολλές χώρες της Ευρωζώνης για τους προπολογισμούς τους τουλάχιστον έχουν λάβει απόφαση μείωσης της φορολόγησης της εργασίας ιδίως για τους πτωχότερους. Η Γαλλία, η Λετωνία και η Εσθονία είναι τέτοια παραδείγματα. Τώρα για τις δαπάνες στους προϋπολογισμούς. Οι διορθώσεις του τα προηγούμενα χρόνια ήταν τεράστιες που χρειάζονταν. Και επίσης έχει σημειωθεί μεγάλη μείωση των δημοσίων δαπανών. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό συνέβαλε σε ανάπτυξη, αλλά χρειάζονταν δραστικές αποφάσεις για τη διόρθωση των προϋπολογισμών. Το 14 και τώρα αρχές 15 τα σχέδια προϋπολογισμών των χωρών μελών δείχνουν ότι περαιτέρω μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες δεν έχουν ζητηθεί. Πρέπει λοιπόν να γίνεται μια συνεχής αναθεώρηση και εξέταση των προϋπολογισμών των χωρών μελών και αυτό έχει γίνει για πολλές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Δανία, την Ισπανία, την Σουηδία. Τα συμπαράσματα δε από αυτές τις αναλύσεις είναι θετικά για τη γενική δημοσιονομική διαχείριση ή διακυβέρνηση της Ένωσης. Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη πρέπει να τονίσουμε τι μέτρα προ... πρότειναν τα θεσμικά όργανα για περαιτέρω στήριξη των μεμονωμένων προσπαθειών κρατών μελών ώστε να τα οθήσουν να διορθώσουν τα ελλείμματά τους, τα δημοσιονομικά τους. Έγιναν ανακοινώσεις για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για τα, μέτρα, τα αντισταθμιστικά μέτρα της ΕΚΤ. Τέλος, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης είναι το κοινό μας σχέδιο. Δεν αρκεί μόνο να αναφέρουμε συνθήματα και κανόνες πρέπει τελικά να δούμε στην πράξη ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να μας ωφελεί όλους, ακόμη και αν μερικές αποφάσεις είναι δύσκολες και σκληρές στην αρχή, μπορεί τελικά να καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα. Για την εφαρμογή λοιπόν της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής Μπορεί να χρειαστεί να παραδώσουμε ένα τμήμα της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος να οικοδομήσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον. Ευχαριστώ. And now I would like to give a floor to Mr. Mr. Ευχαριστούμε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Όλι Ρεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά μαζί σας για να συζητήσω τα πιθανά επόμενα βήματα της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων. Θα ξεκινήσω εκτιμώντας το που βρισκόμαστε σήμερα. Εφτά χρόνια μετά από την αρχή της οικονομικής κρίσης και πέντε χρόνια μετά από την κρίση χρέους που χτύπησε την Ευρώπη πολύ σκληρά. Η σταθεροποίηση από το 2010 μέχρι το 2012 ήταν ε, ικανή να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακάμψει από την άνοιξη του 2013. Αυτό όμως ε, εξασθένισε τελικά τους ρυθμούς ανάπτυξης και η ανεργία έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες της Ένωσης, σαν και σε κάποιες άλλες, βλέπουμε ότι έχει υπάρξει μια βελτίωση. Η ορίμανση ουσιαστικά των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε σε πολλές οικονομίες να επιστρέψουν στην ανάπτυξη το 13 με 2014 αλλά μια συνολική ισχυρή αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη δεν υπήρξε ουσιαστικά στις χώρες της Ένωσης. Και κάποιες γεωπολιτικές εντάσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ και το θέμα του Ισλαμικού κράτους, όλα αυτά οδήγησαν τελικά σε ένα αποπληθωρισμό και σε μία περίοδο ε, ακόμα μεγαλύτερης μείωσης των πληθωριστικών τάσεων. Αυτό υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των οικονομικών εταίρων και εξασθένησε γενικότερα την οικονομική ανάκαμψη, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο έτος. Πιο πρόσφατα υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες επηρέασαν το οικονομικό τοπίο στην Ευρώπη. ανοίγοντας κάποιες καλύτερες προοπτικές. Καταρχάς η δραματική μείωση της τιμής του πετρελαίου έχει επηρεάσει γενικότερα τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Δεύτερον, το λεγόμενο quantitative easing. Αυτή η πολιτική ήταν ουσιαστικότερη από αυτή που πιθανώς θα περίμεναν οι αγορές και ήταν ακριβώς το ισχυρό όπλο το οποίο θα οδηγήσει στην ανάκαψη της Ευρωζώνης. Και τέλος και η οικονομική, αμερικανική συγγνώμη, οικονομία έχει εξελιχθεί και αναπτυχθεί πολύ θετικά και έχει δημιουργήσει θετικές ε, εξελίξεις και για την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκυρία αυτή. Οι αλλαγές αυτές είναι αλήθεια, θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή μας κρατούν μακριά από ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά η κάλυψη αυτών των συγκεκριμένων θα έλεγα πεδίων δεν αρκεί από μόνη της. Υπενθυμίζω ότι ο Μπενουά Κερέ, εξαιρετικός οικονομολόγος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφέρθηκε στην παγίδα της προσωποπαγούς οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συνολικές αποτελεσματικές δράσεις, συλλογικές δράσεις, κινδυνεύουμε εμείς να πέσουμε στην παγίδα αυτή. Με διαρθρωτικά επίπεδα, έμονα επίπεδα ε, θα έλεγα υψηλά ανεργίας, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει γενικότερα και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Τώρα, μπορεί η Ευρωζώνη να διαφύγει από αυτή την παγίδα της προσωποπαγούς ε, οικονομίας και μπορεί να περάσει σε ένα ευρύτερο σχήμα το οποίο χρειάζονται σήμερα ε, οι νέοι της Ευρώπης. Βραχυπρόθεσμα, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου δημιουργούν καλές πρόπτικες για την Ευρώπη. Μέσο πρόθεσμα όμως και μάκρο πρόθεσμα απαιτούνται και περαιτέρω ενέργειες και δεν απαιτείται μόνο ανάληψη δράσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναγνωρίζω την περιπλοκότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Όμως τελικά πρέπει να πούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν την μεγάλη ευθύνη και τις περισσότερες αρμοδιότητες. Η ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι χαμηλές τιμές των καυσίμων μπορούν να επηρεάσουν θετικά, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και τα περισσότερα αυτά πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απαιτείται καλύτερη πολιτική μορφή συντονισμού στην Ευρώπη. Υπάρχουν αρκετές χώρες, μεγάλες χώρες της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας που επηρεάζουν ε, ιδιαιτέρως την οικονομική ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία επιπλέον σημεία. Πέραν δηλαδή της δράσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Νομίζω ότι έχουμε πολλά μέτωπα να καλύψουμε. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το άλλο είναι να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Αυτό απαιτείται όχι μόνο στην Ιταλία και στη Γαλλία. Έτσι ώστε η ποσοτική χαλάρωση να γίνει ιδιαιτέρως αποτελεσματική και να φτάσει στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά. Αυτό είναι σημαντικό και για άλλες χώρες μικρότερες όπως η Φιλανδία, οι οποίες για πάρα πολύ καιρό έχουν καθυστερήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και πληρώνουν σήμερα το υψηλό κόστος της απώλειας ανταγωνιστικότητας και αυξημένης ανεργίας. Εν τω μεταξύ η Γερμανία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον μεγάλο, τον τεράστιο ε, δημοσιονομικό της περιθώριο, το τεράστιο δημοσιονομικό της δυναμικό για να ενισχύσει γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία και τα πλεονάσματά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να οδηγήσουν στην επιτυχία της προσπάθεια του στρατηγικού προγράμματος των 315 δισεκατομμυρίων. Να μην μείνει ε, γράμμα κενό, άνευ περιεχομένου η προσπάθεια αυτή και να ωφεληθεί και η πράσινη ανάπτυξη ε, και γενικότερα η οικονομική δραστηριότητα ευρύτερα. Αυτές είναι προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Πρώτον λοιπόν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να δώσει νομισματικά κίνητρα ουσιαστικά. Δεύτερον, οι χώρες θα πρέπει να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις τους για να προωθήσουν τη δημοσιονομική τους ανταγωνιστικότητα και οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα πλεονάσματά τους και να ευνοήσουν επίσης όλες οι χώρες και την αύξηση των επενδύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές, σε σχέση με την εφαρμογή του συμφώνου, δεν υπάρχει μία ενιαία λύση, δεν υπάρχει μία ενιαία συνταγή για όλους. Γιατί κάθε χώρα έχει ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας. Οι κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί φυσικά, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοούμε και την ευελιξία, η οποία θα πρέπει να υπάρχει και να εφαρμόγεται. Σε σχέση με τις βαχυπρόθεσμες προσπάθειες αποκατάστασης της ισορροπίας, έχουμε τα λεγόμενα εκ των προτέρων ρυθμιζόμενα προγράμματα, τα οποία θα λειτουργήσουν σαν αναφορά ε, σε ορισμένα Έχουμε το παράδειγμα ότι η Ιρλανδία το 2015 προβλέπεται να έχει 3,5% και άλλες χώρες πάνω από 3%. Πολλές χώρες έχουν δείξει ότι οι δημοσιονομικές από τη μία προσπάθειες εξυγίανσης και οι μεταρρυθμίσεις από την άλλη μπορεί να βοηθήσουν έτσι ώστε να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Υπάρχουν τρία επιπλέον στοιχεία τα οποία νομίζω είναι απαραίτητα για μια σταθερή και ουσιαστική ανάκαμψη στην Ευρώπη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρώτον, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια πραγματικά παρεμβατική νομισματική πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Δεύτερον, απαιτείται μια συνεχής προσπάθεια εξυγίανση των δημοσιονομικών των κρατών μελών. Και τρίτον, Απαιτείται η εντατικοποίηση των διαφθορτικών αλλαγών έτσι ώστε η Ευρώπη να καταστεί πιο καινοτόμος, πιο ανταγωνιστική και πιο ευέλικτη. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη βγήκε από την εντατική θεραπεία. Όμως έχουμε ακόμα προσπάθεια να κάνουμε. Πρέπει να νικήσουμε την κρίση και να ισορροπήσουμε την κατάσταση μετά από τις μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί το ίδιο το οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο. Δεν μπορούμε να εμείνουμε στο status quo, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μία μόνιμη παρακμή και δεν θα πρέπει από την άλλη να διαλύσουμε και το ευρωπαϊκό πρότυπο. Γιατί νομίζω ότι και η κοινωνική δικαιοσύνη και η επιχειρηματικότητα οφείλουν πολλά στο ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Σας ευχαριστώ κύριε Ερέν. Τώρα εσείς κύριε Ντόμινικ Χάνεγκαν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι που βρήκατε, μπορέσατε να βρείτε ευκαιρία να παρέμβετε στην συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ και μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ και μπορώ να σας απευθύνω το λόγο για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Θα αναφερθώ πρώτα στο Ιρλανδικό περιβάλλον. Όμως νομίζω ότι τα διδάγματα που αντλήσαμε από εκεί μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες αν όχι όλες τις χώρες μέλη. Τρία χρόνια τώρα έχουν περάσει από τότε που ψήφισαν οι Ιρλανδοί σε εθνικό δημοψήφισμα για να ακυρώσει η Ιρλανδία το δημοσιονομικό σύμφωνο και δύο χρόνια από τότε που άρχισε να ισχύει τον Ιανουάριο του 2013. Θεώρηθηκε τότε ότι ήταν ο πρώτος θεμέλιος λήθος για μια νέα δημοσιονομική ένωση. Τώρα τρία χρόνια μετά, ίσως είναι ακόμα νωρί για να κρίνει κανείς τελεσίδικα το Fiscal Compact, διότι ακόμα ορισμένες χώρες μέλη προσπαθούν να ελέγξουν τα επίπεδα χρέους και ελλείμματος. Όμως, είναι μια συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί για δύο λόγους. Πρώτον, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο υποτίθεται θα ενσωματωθεί στο βασικό σώμα των κανόνων της Ένωσης, στην βασική νομοθεσία της Ένωσης και αυτό χρειάζεται χρόνο και πολλή προετοιμασία. Δεύτερο είναι σαφές ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για ορισμένες χώρες μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο και μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέπει. Το Fiscal Compact επίσης απαιτεί και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου. Έχουμε εμεί το, ανάλογο όργανο στην Ιρλανδία και το έχουμε δώσει και κάποιους ρόλους. Δηλαδή εξετάζει τις προγνώσεις της κυβέρνησης, το που ε, βρίσκεται, παρακολουθεί και αξιολογεί την συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και αξιολογεί εάν η αδίποτε μη συμμόρφωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ με κάποια ικανοποίηση να πω ότι έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που από το Fiscal Compact και ας μην λησμονούμε ότι βασικός του στόχος είναι η σφυριλάτηση μιας μακροχρόνιας, μιας μακροπρόθεσμης δηλαδή, δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το ερώτημα είναι θα μπορέσει να γίνει αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα υπάρχουν και πολύ σημαντικά δημόσια χρέη στις, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμούμεθα όλοι ότι η έγκριση του Fiscal Compact έγινε μετά από την έγκριση μέτρων από το 2008 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μέτρα ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, νομοθετικά και άλλα μέτρα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και διάφορα άλλα όργανα επίγουσας χρηματοδότησης. Πολλές από τις διατάξεις του Fiscal Compact καλύπτονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις μετά από το ξέσπασμα της κρίσης, το ΣΥΚΣΠΑΚ για παράδειγμα και το ΤΟΥΠΑΚ και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο καλύπτουν πολλά από τα όσα ήδη περιλαμβάνονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Η πιο σημαντική καινοτομία του Fiscal Compact ήταν η θέσπιση του χρυσού κανόνος που βάζει ως στόχο εξυγίανση των προϋπολογισμών. Βέβαια αυτό είναι περίπλοκο και το συζητούν ακόμη και οι καλύτεροι οικονομολόγοι μας και δεν έχουν συμφωνήσει πάνω σε μια μέθοδο για να τηρηθούν οι δημοσιονομικές ισορροπίες. Να λοιπόν η αβεβαιότητα που έχει ε, προκύψει από την διαδικασία αυτή και οι σημαντικές προσπάθειες που χρειάζεται για να επιτευθούν οι ισορροπίες. Αβεβαιότητα που ωστόσο ίσως οδηγεί και σε μια έλλειψη προσπαθειών να επιτευθούν οι στόχοι ή μικρότερες από τις αναγκαίες διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι αναποτελεσματικό. Χρειάζεται όμω ξεκάθαρο ορισμός λιγότερο περίπλοκων κανόνων, καθώς επίσης και μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που θεσπίζει. Όπως και τα άλλα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιρλανδία συμμετέχει στο SGP και βεβαίως και λόγω της χρηματοπιστωτικής μας κρίσης ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το διορθωτικό σκέλος με διαδικασία για μείωση του ελλείμματος για να επιστρέψει η χώρα σε βιώσιμες δημοσιονομικές πολιτικές. Τα καλά νέα για την Ιρλανδία είναι ότι πορευόμαστε καλά για να μειώσουμε το ε, υπερβάλλον έλλειμμα μέχρι τα τέλη του 2015 και μετά τα δημόσια οικονομικά της Ιρλανδίας θα μπουν πλέον στο προληπτικό, στο σκέλος πρόληψης και όχι στο διορθωτικό. Το οποίο σκέλος πρόληψης προβλέπει και ετήσια διόρθωση χωρίς να διευκρινίζει πότε θα πρέπει να λαμβάνεται αυτή η θέση. Όταν μπήκαμε στο, θα μπούμε στο, στο σκέλος πρόληψης θα εξετάζεται και το αν συμμορφωνόμαστε προς το ε, δημοσιονομικό benchmark Και βεβαίως έχουμε το όριο των 0,5% ανά χρόνο. Υπάρχει και ένας κανόνας που λέει ότι για παραπάνω από 60% του ΑΕΠ θα πρέπει να μειώνεται κατά ένα εικοστό τουλάχιστον τον χρόνο και προβλέπεται μεταβατική περίοδο για χώρες μέλη όπως η Ιρλανδία που έχει περάσει από διαδικασία ε, ε, υπερβολικού, ελλείμματος από τον Νέμβριο του 2009 και αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2019 δεν θα ισχύει αυτός ο κανόνας του ενός εικοστού. Θα έπρεπε όμως μέχρι τότε να έχουμε κατέβει από το 123% που από δύο χρόνια σε περίπου 90% του ΑΕΠ μας. Δηλαδή θα φτάσουμε να κατεβαίνουμε κατά το 1,5% πλέον από εκεί κάθε χρόνο. Συμπληρωματικά τώρα υπάρχει και ο κανόνας του οροσίμου των δημόσιων δαπανών που θεσπίζει και τη χρηματοδότηση των διαφόρων Υπουργείων. Και αυτό με μια πολύ αυστηρή φόρμουλα και οποιασδήποτε επιπλέον επιπλέον απαιτήσει των Υπουργείων θα πρέπει να θεμελιώνονται σε συγκεκριμένες προτάσεις αύξησης φόρων. Εάν η Ιρλανδία είχε ακολουθήσει τους κανόνες αυτούς πριν από την κρίση, θα είχε συμβάλει αυτό στο να ξεπεράσουμε ορισμένε από τι βαθύτερε δυσκολίε τι οποίε περάσαμε και βεβαίω και από τι πιο επώδυνε προσαρμογέ που χρειάστηκε να υποστούν οι Ιρλανδοί πολίτε. Οι προσαρμογέ που κάναμε απαιτούνταν για πολλού και διάφορου λόγου. Αφενό βέβαια και λόγω των υποχρεώσεων μα που απορρέουν από το Fiscal Compact, αλλά και λόγω του ότι μειώθηκαν συμπατικά τα φορολογικά μα έσοδα και χρειάστηκε και μια τεράστια διάσωση των τραπεζών που χρειάστηκε να χρηματοδοτήσουν οι Ιρλανδοί φορολογούμενοι. Τώρα και μερικά παραδείγματα της, ε, του ότι μειώσαμε τις θέσεις δημοσιόρης υπαλλήλων κατά 10% τις απολαβές τους μέχρι και 27% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και ως αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες υπέστησαν τεράστια πίεση στην Ιρλανδία. Από τότε βέβαια έχουμε διευρύνει και τη φορολογική βάση βάζοντας και φόρο επί της ιδιοκτησίας, επί της ε, ε, παροχής νερού και άλλους φόρους. Και αυτό που σήμανε τελικά ήταν ότι η Ιρλανδία έβαλε το χέρι στην τσέπη και του τελευταίου Ιρλανδού και του πήρε λεφτά. Το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών είναι ότι η κοινωνική συνοχή στην Ιρλανδία αντιμετώπισε σοβαρότατα προβλήματα. Και σας μιλώ γνωρίζοντας το θέμα και γνωρίζοντα, έχω μιλήσει, μιλήσει και με ορισμένου Ιρλανδού συναδέλφου μου εδώ, υπήρξαμε πολύ τυχεροί στην Ιρλανδία διότι ο Ιρλανδικό λαό αντελήφθη ότι πρέπει να τακτοποιήσει τα του οίκου του. Υπάρχουν όμω άλλε χώρε όπου οι πολίτε δεν αντέχουν άλλο και γι' αυτό χαιρόμαι που βλέπω ότι ο στόχο τη νέα ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να μετατοπίζεται και δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη, στι δουλειέ και στην επένδυση. Εμεί περάσαμε τη δυσκολία και τώρα έχουμε ε, αρχίσει να ελέγχουμε πλέον τις δημόσιες επενδύσεις. Η ανεργία μας έχει κατέλθει από το 15% στο 10%. Εξακολουθεί και είναι πολύ ψηλή. Βάλαμε νέα απασχόληση στο σύστημα και έχουμε μάλιστα εισαγάγει και μειώσει των φόρων. Και όπως είπε προηγουμένως η οικονομική μας ανάπτυξη θα πρέπει να φτάσει μέχρι σχεδόν το 4%. Άρα πιο μακροπρόθεσμα όταν θα ξαναβούμε στο σωστό μονοπάτι του NTO θα είναι πολύ ευκολότερο να σεβαστούμε και τους κανόνες του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Αυτές είναι οι πρώτες μου σκέψεις για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εφαρμογή του Fiscal Compact. Και η συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα εδώ αποτελεί το προϊόν μιας καινοτομίας του Δημοσιονομικού Συμφώνου που ξεκίνησε με διακοινοβουλευτική διαδικασία. Την ρίτα του άρθρου 13, το οποίο άρθρο 13 σημαίνει ότι οι χώρες μέλη μπορούν να συνέρχονται σήμερα εδώ, να συζητούν σε βάθος τα αποτελέσματα όπως ε, της οικονομικής σταθερότητας κλπ. Και με μεγάλη ανυπομονησία αναμένω να ακούσω τις απόψεις και των άλλων απεσταλμένων σήμερα εδώ. Well, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάνακεν. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, συζήτηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο για την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, πώς θα ζητάτε το λόγο δηλαδή. Προσπαθούμε να δώσουμε σε όλους το λόγο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Προκειμένου η διαδικασία να είναι πιο απλή και ο καθένας να ξέρει τι τον περιμένει. Να ξέρετε ότι έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή παρεμβάσεις. Αν θέλετε το λόγο, χρησιμοποιήστε την κάρτα που έχετε μπροστά σας, συμπληρώστε την και δώστε την σε κάποιο κλητήρα. Αυτό ισχύει τόσο για τους εθνικούς βουλευτές όσο και για τους ευρωβουλευτές. Προς το παρόν από τους ευρωβουλευτές δεν βλέπω κάποια αίτηση. Μπορείτε και εσείς να αισθήσετε το λόγο αν θέλετε. Θα δώσω το λόγο πρώτα σε τρεις βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο σε έναν Ευρωβουλευτή, εφόσον κάποιος ζητήσει το λόγο μέχρι τότε. Μετά από τρεις-τέσσερις περίπου παρεμβάσεις θα δίνουμε το λόγο στο πάνελ μας, στους προσκεκλημένους μας εδώ, στους κύριους ομιλητές μας για να σχολιάσουν, να απαντήσουν. Δέχεστε αυτή τη διαδικασία. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Συνεπώς, συνάδελφοι, πρώτος είναι από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, Μάρτα Πίντο. Και μετά, να ετοιμαστεί ο επόμενος, Σανσουρέσκας από την Λιθουανία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Πίντο. Ευχαριστώ. Η Πορτογαλία, όπως ξέρετε, το 2014 βγήκε από το πρόγραμμά της. Με 1% ανάπτυξη εκείνη τη χρονιά Πιστεύω ότι θα πετύχουμε το 3% έλλειμμα σύντομα. Στηριχτήκαμε και μέσα και ε, από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Η Γερμανία βέβαια με μεγάλα πλονάσματα θα έπρεπε να επενδύει περισσότερο. στην ενέργεια, για παράδειγμα, τις διασυνδέσεις. Είναι πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για μας, για να συνδεθούμε ακριβώς με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Οι κανόνες, οι κανόνες δηλαδή του πλαισίου διακυβέρνηση θα έπρεπε να ισχύουν για όλες τις χώρες μέλη. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό τώρα. Καμία χώρα μέλος βέβαια δεν θα πρέπει να φεθεί στην τύχη της όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να δείξουν βούληση οι ίδιες, να αναλάβουν δηλαδή τα βήματα που πρέπει για να πληρώσουν το χρέος τους, για να υπάρξει η δημοσιονομική εξυγίανση. Η πολιτική των χωρών μελών δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς χρειάζονται προσπάθειες από όλες τις χώρες και από αυτές που χρειάστηκε να κάνουν δύσκολες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις. Κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα χρειάζονται επιγόντως βοήθεια, αλλά οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Οπότε δεν θέλουμε ειδική μεταχείριση επειδή μία χώρα θέλει κάτι διαφορετικό και έτσι κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοδόμημα. Οι στόχοι του Δημοσιονομικού Συμφώνου έχουν αποτελέσει αντικείμενο συνένεση σε πολλές χώρες. Με μακροχρόνιες ε, συμφωνίες μεταξύ των μεγαλύτερων, τουλάχιστον αυτό έγινε στην Πορτογαλία, των μεγαλύτερων κομμάτων, και έτσι είχαμε και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να τηρηθούν αυτοί οι στόχοι και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κύριος Ζασουρίνσκας έχει τώρα το λόγο και στη συνέχεια ο κύριος Μπακμαν, Γερμανία. Ο κύριος Ζασουρίνσκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα το θέμα αυτό του Δημοσιονομικού Συμφώνου να το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Εμείς επικυρώσαμε την σχετική συμφωνία το 2012. Στη Λιθουανία άρχισε να ισχύει το 2015, όταν δηλαδή ενταχθήκαμε στην Ευρωζώνη κι εμείς. Για να προετοιμαστούμε, το κοινοβούλιο μας τροποποίησε την νομοθεσία μας ανάλογα και το κράτος, τα εποπτικά όργανα, τα ελεκτικά όργανα ανέλαβαν το καθήκον δημοσιονομικής εποπτείας. Κάτι που άρχισε δηλαδή το 2015. Ξέρουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Είναι να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά ε, νομικά συστήματα θα ενσωματώσουν τα κοινοτικά, όσα χρειάζεται για να μπορούμε και εμείς να είμαστε στην Ευρωζώνη. Το σύμφωνο λοιπόν το δημοσιονομικό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν υπάρχει βούληση να εφαρμοστεί. Υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μερικές χώρες μέλη δηλαδή, οι οποίοι με ελαστικότητα ή φιλελεύθερα ερμήνευσαν και ενσωμάτωσαν στην νομοθεσία του τους κανόνες του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Τι γίνεται με παράλογες υπερβολικές δαπάνες. Η Λιθουανία κατάφερε να βγει από την κρίση κάνοντας τις προσπάθειες που έπρεπε, βέβαια, με τη τίμημα. Υιοθετήσαμε όμως τους κανόνες και τους εφαρμόσαμε. Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ο τελικός στόχος. Πώς να διασφαλίσουμε όμως ότι οι πολίτες μας θα ζουν και καλύτερα. κριτήρια όπως είναι το επίπεδο των μισθών ή άλλοι δείκτες που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ζωής σε μια χώρα, στη Λιθουανία πρέπει να ξέρετε ότι είναι χαμηλή. Ποιος είναι λοιπόν ο δρόμος για τη συνέχεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο επόμενος είναι ο κύριος Τράκμαν, Γερμανία. Και να προετοιμάζεται ο κύριος Καβρίτα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Παρακαλούμε. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Δεν είναι τυχαίο ότι προσπαθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε μία κρίση στην Ευρώπη από τη στιγμή που κάποιες χώρες με υψηλό χρέος συνάντησαν και υψηλότατα επίπεδα ανεργίας. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφθρωτικές πολιτικές οδήγησαν την απόλυτη ανάγκη για εφαρμογή του συμφώνου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ανάκαμψης των οικονομιών. Και στις χώρες των προγραμμάτων οφείλουμε ε, σεβασμό γιατί πέρασαν από δύσκολες συμπληγάδες και από τις ε, δύσκολες αυτές καταστάσεις πρόκειψαν σημαντικές δυσχέρειες και στην Ευρωζώνη και στις ίδιες τις χώρες Ωστόσο τώρα αρχίζουν και παίρνουν την πορεία προς τα πάνω, ε, μάλλον έχουν ξεπεράσει τα δύσκολα. Ακόμα και η ανεργία μειώνεται. Πρέπει όμως να προσέξουμε να μην δράσουμε αντιφατικά. Αφενός συζητούμε εδώ μη συμβατικά νομισματικά μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να αυξήσει τα επιτόκια και να ανεβάσει τον πληθωρισμό μέχρι τα 2 περίπου της 100. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους επενδυτές, να τους προσφέρουμε κίνητρα δηλαδή για να επενδύσουν, εκμεταλλευόμενοι ακριβώ τα χαμηλά επιτόκια. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, διότι πρέπει να υποστηρίξουμε το σχέδιο επενδύσεων του Πρόεδρου Γιούνκερ, αλλά προσοχή να μην προκληθούν νέα δημόσια χρέη. Τις επενδύσεις να τις κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Γερμανία. Άλλωστε ενθαρρύνω τον Πορτογάλο συνάδελφό μου να εξετάσει και τη γερμανική περίπτωση διότι ήδη φτάσαμε να γράφουμε μαύρους αριθμούς το 2014 και θέλουμε να συνεχίσουμε και το 2015 συνεχίζουμε να επενδύουμε για, ήδη από το φθινόπωρο καταθέσαμε πρόγραμμα επενδύσεων της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων και αρχίζουμε τώρα να συζητούμε νέο σχέδιο επενδύσεων τα κάνουμε όμως αυτά διότι δεν αναλαμβάνουμε επιπλέον χρέος Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Ευχαριστούμε κύριε Μπράκμαν. Ο κύριος Καπρίτα τώρα, Πορτογαλία. Και να προετοιμάσει το κύριο Σκράινεμα από την Αυστρία, παρακαλώ. Κύριε Καμπρίτα, έχετε το λόγο. Να σας... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη λύπη μου για την απουσία του Προέδρου του Ευρω... της Ευρωζώνης του κυρίου Ντάισελμπλουμ γιατί θα ήταν καλή μια συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε την ανάγκη να σκεφτούμε να αναλύσουμε τις ελλείψεις αυτού του δημοσιονομικού συμφώνου το οποίο δεν ήταν επαρκής ανταπόκριση στη βαθιά κρίση που αντιμετωπίσαμε ούτε ανταπόκριση και απάντηση στην ανάγκη ανάπτυξης και προτεραιότητας στην απασχόληση. Είναι πολύ θετικό που βλέπουμε τις τελευταίες αλλαγές στην ευρωπαϊκή δυναμική νέες αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας και την πολιτική ποσοτικής ελάφρυνσης. Όλα αυτά είναι ουσιώδη για να μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις, να δοθούν βέβαια προτεραιότητες για τις επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες και να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή οικονομία. Τρίτον, μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευληγησία του συμφώνου χρειάζεται. Δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό θέμα το χρέος. Οι 19 χώρες της Ευρωζώνης έχουν όλες μεγάλο δημόσιο έλλειμμα άνω του 90% του ΑΕΠ και η στρατηγική της λιτότητας υπό την προηγούμενη Κομισιόν εμβάθυνε την κρίση και χειροτέρεψε την ύφεση. Η Ευρώπη λοιπόν βρίσκεται σε στασιμότητα και στα πρόθυρα του αποπληθωρισμού. Η Πορτογαλία είναι καλό παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα της Τρόικας που ελπίζουμε να σταματήσουν γιατί δεν έχουν δημοκρατική νομιμότητα έδειξε ότι μειώθηκε η ανταγωνιστικότητά μας και σήμερα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει δυσκολίες που δεν γνωρίζαμε πριν από τρία χρόνια μόλις. Η συνέπεια, η συνοχή λοιπόν του ευρωπαϊκού οράματος, το μέλλον του, περνάει από την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην καινοτομία και στις επενδύσεις με ευρύ περιθώριο ελιγμών και για προλήψεις των κρίσεων και για τις χώρες ιδιαίτερα που υφίστανται τα διορθωτικά μέτρα έστε να μπορούν να γίνουν προσαρμογές για την αντιμετώπιση του χρέους και του ελλείμματος. Να λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικοί κύκλοι, γιατί χωρίς αυτά δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην πλήρη απασχόληση. Ευχαριστώ και ακολουθεί ο κύριος Κράινερ από την Αυστρία. και μετά θα ακολουθήσει ο Ιταλός κ. Γκουαλτιέρη. Κύριε Κράινερ, έχετε το λόγο κύριε. Στα αγγλικά, ευχαριστώ. Ο Όλι Ρεν τόνισε ότι οι ΗΠΑ Πολιτείε βγήκαν από την κρίση ισχυρότερε και τα καταφέρνουν καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέφτει η ανεργία τους, αυξάνει η απασχόλησή τους, πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν διαρωτώμεθα ποια είναι η διαφορά μεταξύ ε, Ενωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως έχουν πολλές αλλαγές και πολιτιστικές και διαφορετικές, πολλές ε, διαφορές θέλω να πω, αλλά ποια είναι η διαφορά στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική που άσκησαν. Νομίζω ότι οι διαφορές τους είναι κυρίως στις προτεραιότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ενωμένες Πολιτείες είχαμε παρόμοιους στόχους για την αναχρηματοδότηση του δημοσιονομικού συστήματος και των τραπεζών κτλ. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν εμεί θέλουμε δουλειέ, απασχόληση, ξεχάστε το έλλειμμα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ακριβώ το αντίθετο. Είπαμε ότι το έλλειμμα και η μείωσή του είναι το πιο σημαντικό. Α ξεχάσουμε και την ανάπτυξη, α ξεχάσουμε και τι δουλειέ. Κάναμε λάθο. Πήραμε τη λάθο απόφαση. Φαίνεται πως οι Ηνωμένες έβαλαν σωστές προτεραιότητες. Άρα λοιπόν πρέπει να ξανασκεφτούμε τις προτεραιότητες μας γιατί αυτές που έχουμε τώρα αποδείχτηκαν λάθος. Δεύτερο, μιλάμε πάντα για ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε λόγο που ακούμε κάποιος λέει ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα. Βέβαια αυτό έχει σχέση με την ελεύθερη οικονομία της αγοράς και βεβαίως μια, οικονομία, μια ε, ανταγωνιστικότητα δεν έχει σχέση με την πολιτική. Εγώ δεν έχω μια ανταγωνιστικότητα απέναντι σε κανέναν από εσά. Άρα, το ισχυρό μα σημείο είναι η συνεργασία, όχι η ανταγωνιστικότητα. Αν ανταγωνιζόμαστε μεν του δε, ήμασταν, υπήρξαμε, περικόπταμε τους φόρους υπέρ εκείνων που τους ή άλλως είχαν αρκετά μεγάλα εισοδήματα, κυρίως πλούσιους και μεγάλες επιχειρήσεις. Ερώτημα, γιατί να συνεχίσουμε σε αυτό αυτή την οδό της ανταγωνιστικότητας εφόσον αυτό ωφελεί μονάχα το τμήμα εκείνο της κοινωνίας που δεν χρειάζεται βοήθεια. Ενώ αυτοί που χρειάζονται βοήθεια πληρώνουν όλο και υψηλότερους φόρους. Αφού ορισμένοι δεν φαίνονται αλληλεγγύοι. Α σκεφτούμε καλύτερα λοιπόν την συνεργασία, όχι τον ανταγωνισμό. Εγώ βλέπω η ανθρωπότητα να προχωρεί και οι μεγάλες πρόοδοι έγιναν πάντα σε βάση συνεργασίας και όχι σε βάση ανταγωνισμών και ανταγωνιστικότητας να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ο κύριος Γκουεριέρη από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα διάφορες παρεμβάσεις, αρκετά αισιόδοξε για την δυνατότητα η ανάκαμψη αυτή η σημερινή να οδηγήσει σε ένα δρόμο σταθερής ανάπτυξης για την Ευρώπη και το ευρώ. στα πλαίσια της υπόθεσης ότι μια πιο ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων και των αριθμιστικών πολιτικών σε συνδυασμό με τις διαφθορτικές μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια, δεν το αμφισβητώ. Υπήρξαν βελτιώσεις σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες ε, χτυπήθηκαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Να μην ξεχνάμε όμως ότι οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν κυρίως γιατί το σύστημα αυτό, η διαδικασία αυτή, επευλήθη με ασύμετρο τρόπο στις χώρες ε, οι οποίες ε, χρωστούν χρήματα. Οι χώρες οι οποίες δανείσαν χρήματα έχουν συνεισφέρει κατελάχιστον θα έλεγα σε αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας της ζώνης του ευρώ. Αυτή η έλλειψη συμμετρίας με φοβίζει για το μέλλον. Με φοβίζει γιατί στην ουσία αυξάνει τις αποπληθωριστικές τάσεις οι οποίες κυριαρχούν στην παρούσα φάση. Ξέρετε ότι το πρόβλημα των χρεών των περισσότερων από τις χώρες αυτές δεν διορθώθηκε. Εάν πράγματι λοιπόν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά η οικονομία της Ευρωζώνης, έχουμε ανάγκη από ένα πλαίσιο ανάπτυξης ένα πλαίσιο ανάπτυξης το οποίο μπορούν να στηρίξουν και να ευνοήσουν μόνο οι λεγόμενες επεκτατικές πολιτικές. Στην ουσία έχουμε αυτή τη στιγμή πέσει σε μια παγίδα σε σχέση με τη μείωση από τη μία της ζήτησης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την αυξήσουμε και μέσω νομισματικών πολιτικών και μέσω δημοσιονομικών πολιτικών και μέσω επενδυτικών πολιτικών που θα οδηγήσουν στη μεγέθυνση των μεγεθών. Θα πρέπει να, να αλλάξει η κατάσταση, να μην υπάρχει αυτή η ασυνέχεια η οποία χαρακτηρίζει την οικονομία. Το να πιστεύει κανείς ότι κάποιες επιμέρους περιφερειακές ρυθμίσεις ε, θα διορθώσουν τα πάντα είναι λάθος. Αυτό θα προκαλέσει αύξηση του κόστου σε εισαγωγικά επισκευή της οικονομίας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να αγνοήσω και γι' αυτό επιμένω υπογραμμίζοντάς το. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μας για κάποιες σύντομες απαντήσεις. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ράιρς. Σας ευχαριστώ. Όντως έχω κάποια σύντομα σχόλια. Πρώτον, συγχαρητήρια στην Πορτογαλία. Ο Υπουργό Οικονομικών σας είπε ότι είναι έτοιμη η Πορτογαλία να αποπληρώσει τα δάνειά της πριν λήξει προθεσμία στο Διεθνές Μεσματικό Ταμείο αυτό οφείλεται στις διαφορετικές αλλαγές και στη δημοσιονομική πειθαρχία. Ήταν και η μόνη διέξοδος. Ήταν ο μόνος τρόπος για να βγει η Πορτογαλία από την κρίση. Ακολούθησε το πρόγραμμα και κατάφερε πριν την προθεσμία να βγει από αυτό. Πριν από τρία χρόνια ήμουν εδώ ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου μας και τότε σας είχα πει πώς η δημοσιονομική πειθαρχία συμβιβάζεται με τις επενδύσεις. Όντω, και το παράδειγμα της Λετωνίας αυτό δείχνει. Δείχνει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν εμποδίζει τις επενδύσεις. Εμείς ήμασταν σε πρόγραμμα, υιοθετήσαμε δημοσιονομικά μέτρα, δεν περιορίσαμε όμως ποτέ τις δημόσιες επενδύσεις σε διάφορους τομείς. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες τώρα, ένα σχέδιο και το ίδιο προφανώς δεν ταιριάζει σε όλους. Γι' αυτό όμως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε διευκόλυνση. Το Συμβούλιο επίσης πρότεινε κάτι για τις κεφαλαϊκές αγορές και υπάρχει βέβαια και το επενδυτικό σχέδιο Juncker. Οι Υπουργοί Οικονομικών στο ΕΚΟΦΗΝ κατέληξαν ότι το σχέδιο το επενδυτικό Juncker δεν περιορίζεται, είναι κάτι παραπάνω, δεν περιοριζόμαστε δηλαδή σε μεταρρυθμίσεις, διευθυντικές μεταρρυθμίσεις μόνο. Συμπληρώνει την εικόνα το επενδυτικό αυτό πακέτο, αποτελεί ένα παραπάνω μέσο για να βγούμε από την κρίση. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Εξάλλου, το πακέτο Juncker προβλέπει ιδιωτικέ επενδύσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αξιολογήσει τα προγράμματα και μόνο τα προγράμματα εκείνα τα οποία έχουν ω στόχο την αυτοχρηματοδότηση και θα αποφέρουν οι επενδύσεις που θα γίνουν θα εγκριθούν τελικά. Τώρα, όσον αφορά τη φορολογία φορεσοδήματος. Στο Συμβούλιο την τελευταία φορά εγκρίναμε οδηγία όσον αφορά την ανακατανομή του εισοδήματος. Και βάσει αυτής της νομικής πράξης οι φόροι πρέπει να πληρώνονται ε, εκεί όπου έχει λάβει η χώρα οικονομική δραστηριότητα και από όπου προέρχεται δηλαδή το κέρδος. Θέλω να καταλήξω ή να απαντήσω σε μια ερώτηση που άκουσα νωρίτερα. Ακούστηκε πολλές φορές το παράδειγμα της Αμερικής και η ανάπτυξη που έχει τώρα η Αμερική. Θυμηθείτε όμως τι έγινε με το αμερικανικό δολάριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζούμε στην παγκοσμιοποίηση. Και οι οι οικονομικοί κανόνες ισχύουν παντού. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι κανόνες αυτοί μπορούν να αλλάξουν ή να παρακαμφθούν. Η βασική διαφορά όμως ανάμεσα σε εμά και την Αμερικανική οικονομία είναι η εξή. Πρώτον, τα όρια και οι ανισότητες στα εισοδήματα είναι πιο χαμηλές στις χώρες μέλη. 40% του προπολογισμού μας πηγαίνει στην ε, Λετωνία σε κοινωνικές παροχές. Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εμά και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Στις Ηνωμένε Πολιτείες, καλά Αμερική είναι Αμερική βέβαια, αλλά η Ευρώπη προσέχει την κοινωνική προστασία. Θέλει να αποφύγει τις μεγάλες ανισότητες. Μας ενδιαφέρει η ίση κατανομή των ε, εσόδων. Αυτή είναι μια βασική διαφορά στην δικιά μας οικονομία σε σχέση με την Αμερικανική. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε όλοι ε, στο ίδιο βήμα, δηλαδή στον ίδιο βηματισμό, δηλαδή όλοι θέλουμε την ισότητα, όλοι θέλουμε την κοινωνική προστασία και όλοι θέλουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Και θέλουμε βέβαια επιπλέον επενδύσεις και ανάπτυξη. Όχι όμως σε βάρος των κοινωνικών μας κεκτημένων. Ούτε θέλουμε να αποκτήσουμε νέα δάνεια και νέα χρέη. Ο κύριος Ρεν τώρα. Κύριε Ρεν, θέλετε κι εσείς να σχολιάσετε, να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατος γιατί συμφωνώ εν με τον προηγούμενο μιλητή. Για την Πορτογαλία ακούσαμε δύο εξαιρετικές παρεμβάσεις περί αυτής και το βρίσκω ενθαρρυντικό και σημαντικό ότι η Πορτογαλία μαζί με την Ιρλανδία, Ισπανία κατάφεραν να βγουν από το πρόγραμμα στήριξης εγκαίρως ή ακόμη και πριν να λήξει επίσημα και επέστρεψαν στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη καθώς και βελτίωσαν την ε, κατάσταση ως προς την απασχόληση. Οι επίπονες αποφάσεις που είχαν ληφθεί Είχαν βέβαια επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά τώρα αυτά έχουν αποτέλεσμα και αναγνωρίζεται αυτό. Όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα προγράμματα, όντως βοηθάνε τις χώρες να ανακάμψουν. Το είδαμε στην Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω τον κύριο Πίντο ή όπως είπε και ο κύριος Πίντο πρέπει να είναι οι ίδιοι οι κανόνε για όλου μάλιστα. Για τη Λιθουανία που μπήκε στο ευρώ την 1η Ιανουαρίου φέτο θα ήθελα να τη συγχαρώ. Αν θυμάστε η Λετωνία το περασμένο χρόνο και η τρίτη βαλτική χώρα πριν από 2-3 χρόνια αποφάσισαν όλες και οι τρεις βαλτικές χώρες να είναι μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και όπως είδαμε από τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρες αυτές ήταν σωστή η απόφαση τους αυτή γιατί μπόρεσαν να πετύχουν επενδύσεις και σημαντική οικονομική και κοινωνική σταθερότητα που στηρίζουν την ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Για το μέλλον της Τρόικας όπως είπε ο κύριος Καμπρίτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην σχετικά πρόσφατη έκθεσή του, περσινή δηλαδή, για την Τρόικα ενθαρρύνει, συστήνει μία αναθεώρηση της λειτουργίας της Τρόικας και μπορεί να θυμάστε ότι αρχικά στις αρχές του 2010 τα κράτη-μέλη επέμειναν να συμμετάσχει και το Δουνουτού γιατί δεν υπήρχε πλήρης εμπιστοσύνη για, από όλους για την ανεξαρτησία της Κομισιόν και την επαγγελματικότητά της. Μερικοί είχαν αμφιβολίες δηλαδή. Γι' αυτό έγινε η επιλογή να μην τα κάνει όλα η Κομισιόν που έχει δημοκρατική λογοδοσία αλλά να συνεργαστούμε και με το δουνοτού και την ΕΚΤ. Στην ε, αναθεώρηση αυτή η κεντρική ιδέα είναι ότι η δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να ε, τύχει εγγύησης από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Και από την εμπειρία που έχω θα έλεγα ότι και στο μέλλον εφόσον υπάρξουν τέτοιες κρίσεις και χρειαστούν τέτοια προγράμματα προσαρμογή, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θέλουμε για το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Εκτός αυτού πρέπει να δούμε ακόμη αν τα κράτη-μέλη θέλουν να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και από το Δουνουτού γιατί και το Δουνουτού έχει πολύ αυστηρούς κανόνες που προβλέπουν ότι αν χορηγήσει χρηματοδότηση πρέπει να έχει και λόγο για το πρόγραμμα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν υποστηρίζω την εξέταση που έγινε για το ρόλο της Τρόικας και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και μια γενικότερη εξέταση και αναθεώρηση της δημοσιονομικής λειτουργίας της Ευρωζώνης. Καθώς και το ότι η Ευρωζώνη πρέπει να είναι σε θέση να έχει εκπροσώπους ε, και στις συνεδριάσεις με το ΔΝΤ, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης, άρα δεν έπαιξε το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει έναντι του Δουνουτού η Ευρωζώνη. Ενώ αντίθετα αν είχαμε ενώσει τις προσπάθειές μας και στο Z20 και αλλού θα είχαμε πολύ περισσότερο ειδικό βάρος και δεν θα μας τα καθόριζε όλα η ΙΠΑ και η Κίνα αν θέλουμε επαναλαμβάνω να παίξουμε τον πλήρη ρόλο που μπορούμε να παίξουμε διεθνώς στα διεθνή βήματα για οικονομική διακυβέρνηση. Τέλος για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη. Περάσαμε από τη σταθεροποίηση στην επένδυση και την ανάπτυξη, όπως είπε και το πρωί ο Πιέρ Μασκοβισή. Εδώ η Τραπεζική Ένωση Uh, and uh, now we have to continue with... Κατέληξε ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις για να διευκολυνθεί η οικονομική αύξηση και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρέν. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτά που είπατε, ιδιαίτερα τη φράση σας για τον πολιτικό σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Και τώρα θα θέλαμε να απαντήσει ο κύριος Χάνιγκαν. Να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο Πίντο για την Πορτογαλία. Όπως και εμείς περάσαμε από ένα τέτοιο πρόγραμμα, είδαμε ποιοι ήταν οι κανόνες, σεβαστήκαμε τους κανόνες, και θα με ανησυχούσε να υπάρξει ειδική μεταχείριση για κάποιο άλλο κράτος μέλος. Βέβαια καταλαβαίνω τα επίπεδα της κρίσης. Η διαδικασία ρύθμισης δεν αντιμετώπισε γενικά τα προβλήματα του χρέους όπως είπε και ένας συνάδελφος πριν. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει συνολικά, όχι για ένα κράτος μέλος, γιατί αλλιώς θα δούμε μια μετακίνηση από το κέντρο προς τα περιφερειακά κράτη και αντί να λύσουμε το πρόβλημα μια συγκεκριμένη χώρα. θα βλέπουμε ότι οι χώρες θα επανέρχονται και θα ζητούν η κάθε μία μια ειδική μεταχείριση. Αυτό δεν είναι σωστό. Οι χώρες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι σαν ένωση έχουμε κανόνες, είμαστε μια ένωση ποιότητας, μια ένωση δικαιοσύνης και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Thank you very much. And now to share our business, we are switching our chairmanship. Τώρα αλλάζουμε λοιπόν την Προεδρία. Αναλαμβάνει ο κύριος Session. Ο κύριος Γουαλτιέρη. No, I think you can stay here. Yes. Perfect. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Νέπερους από την Ολλανδία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένα σταθερό ευρώ έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις οικονομικές αγορές και την οικονομική θέση της Ευρώπης. Γι' αυτό το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο πολύ, ή μάλλον πολύ σημαντικό γιατί μας κρατάει και σε δυνατή θέση. Παρόλο που χρειάζονται θυσίες, δεν πρέπει αυτό να το αποσιωπούμε. Είναι αλήθεια ότι πολλέ χώρες με τις μεταρρυθμίσει νιώσανε πολύ άσχημα. Δεν πρέπει βέβαια να τους λέμε μόνο ότι πρέπει να κάνετε οικονομίες και ότι πρέπει να κόβετε από κοινωνικές δαπάνες κλπ. κλπ να αυξάνετε τους φόρους. Όλα αυτά πονάνε, κανένας δεν τα αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες και αυτό είναι ανάγκη. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Στην Ευρώπη πρέπει να δράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπανά και πώς. Ως κάτω χώρες και ως κοινοβούλιο των κάτω χωρών περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις προτάσεις για τους ίδιους πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς θα χρηματοδοτείται γιατί είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και τις χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της βέβαια. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μουέ από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Αυστριακός συνάδελφος για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πράγματι βγήκανε γρήγορα από την κρίση του 2009 Ηνωμένε Πολιτείε, εφαρμόζοντας αμέσως μία επεκτατική νομισματική πολιτική και αφήνοντας για αργότερα την δημοσιονομική εξυγίανση. Όταν δηλαδή η Αμερικανική οικονομία είχε επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Στην Ευρώπη δεν το κάναμε αυτό. Δεν το κάναμε γιατί το πρόβλημα της δημοσιονομικής πολιτικής ολόκληρης της Ευρώπης είναι περίπλοκο. Δεν μπορέσαμε να συντονίσουμε τις δημοσιονομικές μας πολιτικές όπως θα έπρεπε. Εξακολουθούσαμε να επιχειρηματολογούμε, η κάθε χώρα να εφαρμόζει τους δικούς της τους κανόνες, χωρίς ποτέ να καθίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα συνολικά. Όταν μια χώρα μπαίνει σε πρόγραμμα εξυγίανσης, μπορεί να αποφεληθεί από την ανάπτυξη των εταίρων της. Άρα μπορεί να κρατήσει ανάπτυξη και να περιορίσει το έλλειμμά της, γιατί στο σύνολο υπάρχει ανάπτυξη και άρα η ύφεση είναι περιορισμένη. Αν όμως όλοι παίρνουν τέτοιου είδους μέτρα, τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε και ως Ευρώπη πρόσφατα, δηλαδή η ύφεση ήταν πάρα πολύ έντονη, γιατί όλοι ακολουθήσαμε τα ίδια μέτρα, μειώσαμε με το διαρθρωτικό έλλειμμα, αλλά από την άλλη μεριά χάσαμε σε έσοδα, φτιάξαμε συγκυριακό έλλειμμα και το είδαμε αυτό. Και μετά μας εκπλήσει που δεν έχουμε ανάπτυξη ή που τελήματα στο σύνολο των χωρών μειώνονται ελάχιστα. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Όπω είπε και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, χρειαζόμαστε ένα πραγματικό συντονισμό των οικονομικών μα πολιτικών, όχι μόνο των δημοσιονομικών. Είναι αναγκαίο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε συγκυριακές καταστάσεις όπως ήταν η κρίση στην οποία βρεθήκαμε. Ευχαριστούμε. Γαλλία πάλι, επόμενος ομιλητής, η κυρία Κέλλερ από τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά, όπως και ο συνάδελφός μου που τόνισε την αλληλεξάρτηση των προγραμμάτων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Γαλλία όπως ξέρετε παρακολουθείται στενά για τα ελλείμματά της και έχουμε συνείδηση της ευθύνης μας ως μεγάλης χώρας για μία από τις κυριότερες οικονομίες της Ευρώπης ότι πρέπει να γίνει μία βιώσιμη και σταθερή διόρθωση του ελλείμματός μας. Πράγμα που καθυστερεί όμως γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της αναδιάρθρωσης της ανεργίας, ε, των κοινωνικών δαπανών, περισσότερο ίσως από ό,τι άλλες χώρες και έχουμε και το πρόβλημα της ακαμψίας της αγοράς εργασίας μας. Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν τη σημασία της νέας ερμηνείας που δίνει η Κομισιόν για την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας που ανακοινώθηκε στις 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό δεν μας αθωώνει δε μας επιτρέπει να παραλείψουμε την προσπάθεια για τη διόρθωση των ελλημάτων και σημειώσαμε στα πρακτικά σημειώσαμε στην ανακοίνωση της Επιτροπής ότι χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και αναλάβαμε τη δέσμευση να το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, για τη λιτότητα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη. Όπως είπαμε και πριν, το σχέδιο Juncker, ας πούμε, είναι σημαντικό, αλλά και η αποτελεσματικότητά του θα είναι σημαντική, αν είναι αποτελεσματικό, για να υπάρξει νέα ανάπτυξη, αλλά και νέα εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, γιατί οι οικονομίες μας αλληλοεξαρτώνται. Για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο αποτελεσματικά, και να καταπολεμηθεί η ανεργία στην Ήπειρό μας. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέσλον από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είχα σκοπό να ζητήσω το λόγο, αλλά αφού πρόκειται αφού μίλησαν οι χώρες της Ευρωζώνης, θα ήθελα και εγώ να πω ότι υποστηρίζουμε αυτά που υπόθηκαν για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Έχουμε πρωθυπουργό που έχει γράψει και ένα βιβλίο σχετικό πρόσφατα και λέει ότι ένα χρεωμένο κράτος δεν είναι ποτέ ελεύθερο. Έχουμε λοιπόν δικούς μας δημοσιονομικούς κανόνες που μας υποχρεώνουν να αποφεύγουμε τα ελλείμματα. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι κάτι που έχει γίνει στη Σουηδία και που θα μπορούσαν να το μιμηθούν και άλλες χώρες είναι ότι η δημοσιονομική μας πολιτική γίνεται σε συγκαθορισμό με τα συνδικάτα και τις επιχειρήσεις για να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά και πιο δίκαια τα μέτρα που προβλέπουμε για να υπάρχει σύνδεση μεταξύ όσων έχουν, διαθέτουν πολλά κεφάλαια και όσων έχουν λιγότερα έτσι ώστε να βγουν όλοι μαζί από την κρίση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει έξυπνη εξοικονόμηση παραδείγματος χάρη αν διαπιστωθεί μεγάλη ανέχεια τότε πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την πραγματικότητα οι δημοσιονομικοί κανόνες. Να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση για, ως προσπάθειες για τη μείωση της ανέχειας αυτής για να μην υπάρξει πτωχοποίηση της οικονομίας μας. Όλοι φυσικά πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους για να μην βλέπουμε πια ανθρώπους να κάνουν ουρά για να τους μοιράζουν σούπα. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν κάποια σύνδεση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής. Και να γίνουν και μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα σύντομα. Δέκα χρόνια είναι πολύ μακρύ διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως η συνθήκη καλύπτει όλα τα συμβαλόμενα μέρη, επομένω και την Σουηδία και η διάσκεψη απευθύνεται και σε χώρες που δεν υπέγραψαν και α, κύρωσαν την ε, συνθήκη, όπως η χώρα του Λόρδου Ντέιβις που ακολουθεί τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Μα δεν έφταιγα εγώ όμως κύριε Πρόεδρε και μάλιστα εγώ προσωπικά εκφράζω τη λύπη μου. Θα ήθελα να πω ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα από όλοι Ρεν και Χάνεγκαν ήταν εντυπωσιακέ και πολύ ενθαρρυντικέ. Αν, εκτός αν ο κύριος Ντάισελ Μπλουμ έχει ενσκύψει τώρα επί του ελληνικού προβλήματος να το λύσει από μόνος του, αν δεν είναι αυτό τότε έκανε λάθος και που δεν ήρθε. Για τα πρώτα χρόνια της κρίσης πάντως θεωρώ ότι υπήρξαν κάποιες προσπάθειες λύσης αλλά και κάποιες ελλείψεις, κάποιες απουσίες και από αυτές έχουν πλήξει κυρίως την Ευρωζώνη και εννοώ την έλλειψη αυτόματου μηχανισμού σταθεροποίησης όπως έχουμε στις επιμέρους χώρες μέλη για παράδειγμα μέσω του συστήματος ε, προστασίας των ανέργων κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ. Και των ποσών που καταβάλλονται δηλαδή είτε από τα συστήματα κοινωνικής ασφαλίσεως, είτε από τους ε, εργοδότες κλπ. Στην περίπτωση ασυμμετρικού αρνητικού σοκ, όπου κάποιες περιφέρειες πλήττονται περισσότερο, αυτοί, αυτές οι περιοχές λαμβάνει αντικυκλικούς πόρους υπό τις περιστάσεις αυτές. Ενώ τέτοιο μηχανισμό δεν έχουμε στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει με απότομο τρόπο. Έχουμε πολύ διαφορετικά επίπεδα επιδομάτων ανεργίας σε διάφορες χώρες μέλη. Θα έπρεπε να έχουμε ένα βασικό ελάχιστο που να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουν οι χώρε μέλη να πηγαίνουν παραπάνω να του επιτρέπεται και βεβαίως και τα επίπεδα διαρθρωτικής ενεργείας στις χώρες μέλη της Ενώσης είναι πολύ διαφορετικά και θα ήταν και λάθος και θα παρήγε το αντίθετο αποτέλεσμα αν οι περιφέρειες εκείνες που έχουν υψηλότερη ενεργεία να επιδοτούν άλλες αλλού. Και ε, επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο ρυθμός αλλαγής της ανεργίας. Νομίζω λοιπόν, με λίγα λόγια, ότι το μέτρο αυτό θα είχε χρησιμότητα αν μπορούσε να θεσπιστεί ένα τέτοιο σύστημα. Και ε, κάπως με απογοητεύει το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί. Thank you. σας ευχαριστώ. Έχει γίνει πρόταση για τον αυτόματο σταθεροποιητή. Θα επανέλθουμε ίσως. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ ε, Λόρδε Ντέιβις για την παρέμβασή σας και θα ακολουθήσει ο κύριος Κέλεμετς από την Εστονική Βουλή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σταματήσουμε τα παράπονα, να σταματήσουμε τη γρίνια και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που βρισκόμαστε όλοι εδώ για να εξετάσουμε από κοινού τους αριθμούς που έχουμε μπροστά μας. Είδαμε ότι οι στόχοι για την Ευρώπη 2020 δεν συνδέονται με την ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους στόχους των επιμέρους χωρών όπως της Φιλανδίας που είναι εξαιρετικοί αριθμοί είναι αλήθεια ότι δεν συνδέεται ε, το επιπλέον έλλειμμα με την ανάπτυξη. Αν και για κάποιους συναδέλφους το βασικό μήνυμα ε, για να υπάρξει ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες δημόσιες δαπάνες. Προτάθηκε επίσης πάρα πολύ σωστά μια πιο προσεκτική εξέταση χωρών όπως η Λετωνία, η Πορτογαλία κτλ όμως και η Δανία, Πολωνία, Σλοβακία, Εσθονία, Τσεχία και αυτές οι χώρες κατάφεραν να προχωρήσουν σε μια διαρκή αηφόρα ανάπτυξη χωρίς επιπλέον δαπάνες. Θα επαναλάβω λοιπόν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σορέν κατά τη διάρκεια της συνάντησης στα πλαίσια της φιλελεύθερης ομάδας. Εάν η επιπλέον δαπάνη σημαίνει ότι θα υπάρξει ανάπτυξη, τότε η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία θα ήταν πρωταθλητές της Ευρώπης σε οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Εφόσον έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να εξετάσετε τους αριθμούς θα καταλάβετε πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ρουμανική Γερουσία η κυρία Κρέτου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι όλες οι χώρες χαρακτηρίζονται με διαφορετικούς βαθμούς ανάπτυξης και με αρκετές οικονομικές διαφορές, μάλιστα και μακροοικονομικές διαφορές. Είναι εφικτή η προσπάθεια να γίνουν βέβαια οι οικονομίες πιο ανταγωνιστικές, αλλά τα μέσα και οι τρόποι δεν είναι οι ίδιοι για τις διάφορες χώρες. Πρέπει να σταθούμε κυρίως στους δείκτες τους οποίους χρησιμοποιούμε και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την πολιτική μας και στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας. Το ΑΕΠ και η εξέλιξη του ΑΕΠ υποτίθεται ήταν το βασικό στοιχείο αναφοράς. Η Ιρλανδία ήταν ηγέτιδα θα έλεγα σε σχέση με τον σεβασμό του κριτηρίου αυτού. Παρά την συγκεκριμένη αυτό όμως συμπεριφορά η Ιρλανδία παρά τα χαμηλά ελλείμματα κατάφερε να είναι ένα από τα κατεξοχήν θύματα της κρίσης. Ζητήθηκε και μία έκθεση για την κατάσταση της οικονομίας έτσι ώστε να κατανοήσουμε γιατί εξεπλάγημεν όλοι από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Ελήφθησαν υπόψη πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αμφισβητούν την κυριαρχία του ΑΕΠ ως κατεξοχήν δίκτυ. Η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση δεν είναι ουσιαστικά αξιολόγηση τομεακή, δεν είναι λεπτομερής. Γιατί χρησιμοποίησαμε ας πούμε το ισοζύγιο πληρωμών αντί για το ΑΕΠ. θα δημιουργήσουμε μια διαφορετική ιεραρχία κριτηρίων. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Από, το, από την Βουλή της Κύπρου ο κύριος Νεοφίτου. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα παράδοξο που το συναντάμε ε, τα τελευταία χρόνια. Η δική μας γενιά διαμαρτύρεται γιατί πρέπει να ήρθε η ώρα που πρέπει να πληρώσουμε τα χρέη που δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Αλλά την ίδια ώρα κάποιοι προτείνουν τη λύση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε για να ξεπεράσουμε τα σημερινά προβλήματα φορτώνοντας το βάρος στις επόμενες γενιές. Δεν θεωρώ πως αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη μιλούμε και στη δική μου χώρα για την αλληλεγγύη που πρέπει η Ευρώπη να επιδεικνύει. Όμως ξεχνούμε ένα άλλο κανόνα. Πέραν της αλληλεγγύης πρέπει να είναι και η δικαιοσύνη. Και δεν είναι δίκαιο άλλοι να δημιουργούν χρέη και άλλοι να τα πληρώνουν. Η ανάπτυξη μέσω επιπρόσθετων χρεών δεν είναι βιώσιμη και πρέπει να επιδιώξουμε την ανάπτυξη μέσα από την δημοσιονομική εξυγίανση. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι αυτή η κρίση μας έδωσε την ευκαιρία να διορθώσουμε ελλείμματα της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Εισήξαμε ένα ευρώ με μόνο κοινή νομισματική πολιτική, εν διαπουσία δημοσιονομικής πολιτικής χωρίς τραπεζική ένωση και χωρίς κοινή εποπτεία. Αυτή η κρίση μας έδωσε την ευκαιρία έστω και αργά να διορθώσουμε λάθη. Θα σχολιάσω τη συζήτηση που γίνεται για το IMF. Δηλαδή θέλουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο τους Ευρωπαίους φορολογούμενους γιατί αν φύγει το IMF η συνεισφορά του πρέπει να αντικατασταθεί από ευρωπαϊκούς φόρους. Και θέλω να πω και την εμπειρία μου από μια χώρα που είμαστε στο πρόγραμμα. Διακρίνω μια σοβαρότητα στο IMF παράλληλα με τη σοβαρότητα των ευρωπαϊκών θεσμών και εμπειρογνωμοσύνη σε συγκεκριμένα θέματα που ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κατά την άποψή μου δρόμο να τα αποκτήσει. Τελειώνω λέγοντας πως ε, η Ευρώπη για να έχει μέλλον οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες. Όσο δύσκολο και αν είναι για κάποιες από εμά τις χώρες πρέπει να μάθουμε να ακολουθούμε τους κανόνες. Οι εξαιρέσει πολλές φορές δημιουργούν και προβλήματα. Thank ε, Uh, Συμπληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο για τις τελικές απαντήσεις στους βασικούς μας ομιλητές. Ο κύριος Ράιευς έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Ναι, μετά από τα προηγούμενα σχολιά μου στον πρώτο γύρο, θέλω να συμπληρώσω μεταξύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κύπριο συνάδελφο που πήρε το λόγο πριν από λίγο. Με ενδιαφέρον να βλέπουμε τις αντιδράσεις και από το κοινό εδώ απέναντι στα θεωρία. Εσείς οι νέοι, κάποιοι από εσά θα χρειαστεί να πληρώσετε τα δικά μας δάνεια. Αλλά Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να τα έχουμε προπληρώσει. Πάντως είναι ενδιαφέρον να ακούσετε τη συζήτηση εδώ για να δείτε τι είδους προβλήματα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε στο μέλλον αν συνεχίσουμε να δρούμε με τέτοιο κοντόφθαλμο τρόπο. Συμφωνώ λοιπόν με τον Κύπριο συνάδελφο και θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είπε και ο κύριος Σντόσκι νωρίτερα όταν σχεδιάζεις με ταπεινό τρόπο τον προϋπολογισμό σου, ε, δεν θέλεις να πρέπει να πληρώνουν τα παιδιά σου, φροντίζεις να πληρώνεις εσύ. Το ίδιο ισχύει και στις χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πρέπει να δούμε πώς θα μειωθεί το βάρος του χρέους. και ό,τι μπορέσουμε να κερδίσουμε πρέπει να το επενδύσουμε ώστε να υποφεληθεί η επόμενη γενιά και όχι να μεταφέρουμε το βάρος στην επόμενη γενιά όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σάνιγκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάποιος από τη Σουηδία είπε πώς βγήκε από την κρίση Σουηδία με τη συνεργασία στην κοινωνία. Στην Ιρλανδία έχουμε μια αντίστοιχη εμπειρία. Δεν ε, θα έλεγα ότι δεν έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση η κοινωνία εξαιτία των μέτρων που υιοθέτησε. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς δεν περάσαμε ούτε μια μέρα με διαδηλώσεις κτλ. Εμείς συζητήσαμε με τους εργαζόμενους, με τους εργοδότες για να αντιληφθούν όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έτσι συνεργαστήκαμε. Ολόκληρη η κοινωνία και η συνεργασία αυτή βοήθησε πολύ. Για αυτά που είπε ο κύριος Νοφίτου, για μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν όπως είναι ο νέος μηχανισμός και, άλλα, και άλλοι μηχανισμοί που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, η ποσοτική χαλάρωση κτλ. γίνονται με συνένεση, όπως και το επενδυτικό πακέτο. Κάνουν πράγματα λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οφελούν, αλλά άκουσα και τον Ντέβι και άλλου ότι υπάρχουν και άλλε προτάσει που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε, αν μη τι άλλο, να μην σταματήσουμε εδώ. Χρειαζόμαστε και συνέχεια. Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε με τίποτα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Όλοι Ρεν. Ευχαριστώ Ρομπέρτο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον τον Ντέιβις για, για αυτά που μας είπε καθώς και τη Βουλή των Λόρδων για όλες τους τις ε, τακτικές εκθέσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία που τις διαβάζω με μεγάλη χαρά και προθυμία γιατί είναι πολύ χρήσιμες. και μας βοηθά να βελτιώσουμε τα προγράμματά μας. Όπως είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν ακουστεί προτάσεις για αυτόματους σταθεροποιητές που είναι θέμα αμφιλεγόμενο στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε τα πράγματα οργανώθηκαν διαφορετικά έτσι ώστε ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός να παραμείνει ψηλός ενώ των μεμονωμένων κρατών να μην έχει έλλειμμα. Και δεν υπάρχει και μηχανισμός διάσωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όλο σύστημα λοιπόν ε, έχει συλληφθεί διαφορετικά. Νομίζω ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες νομίζω ότι οι βασικές κατευθυντήρες γραμμές πρέπει να είναι ότι η αύξηση της αλληλεγγύης πρέπει να πηγαίνει μαζί με μια αύξηση της ευθύνη. Αλληλεγγύη λοιπόν έναντι σταθερότητας. Αυτό είναι η ασχή μας για την οικονομική διακυβέρνηση. Όσο για αυτά που είπαν οι κύριοι Κόλεμετς, που είπε ο κύριος Κόλεμετς, τον ευχαριστώ, διότι και στην Ισπανία υπάρχουν διαφορές που έχει κάνει περισσότερες προσπάθειες από τη Γαλλία και την Ιταλία. Αν σημειώνονται μεγάλα ελλείμματα και αυτό συμβάδιζε με οικονομική ανάπτυξη τότε η Ιταλία και η Γαλλία θα ήταν πρωταθλήτριες της ανάπτυξης και η Φιλανδία για τις βόρειες χώρες αλλά δεν συμβαίνει αυτό και γι' αυτό πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις για την ανάπτυξη, άλλους πόρους από αλλού, ας πούμε επενδύσεις, οικονομικές μεταρρυθμίσεις κλπ. Τέλος προς τον κύριο Μουέ για την νομισματική πολιτική είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και πιστεύω ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε δει μεγάλη εξέλιξη του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης δηλαδή τη μετάβαση από τα LDRO στο OMT και στη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών αγορών. Είδαμε την οικοδόμηση της Τραπεζικής Ένωσης που και αυτή κατέστησε το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα πιο σταθερό και από την καθαρά δημοσιονομική πλευρά είδαμε ενίσχυση της κοινή διακυβέρνησης μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης. Όλα αυτά στις μακροοικονομ... στα μακροοικονομικά προγράμματα έχουν εξισορροπήσει τα πράγματα μεταξύ τραπεζών και η Ευρωζώνη έχει πολύ περισσότερα όπλα αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει καινούργιες κρίσεις πιθανώς στο μέλλον. Με μικρότερο επομένως κοινωνικό και οικονομικό κόστος, ακόμη πιο σημαντικό Ο συντονισμός της πολιτικής στοχεύει στην πρόληψη των κρίσεων και σε σταθερότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει οικονομική διακυβέρνηση. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη διόρθωση εκ των υστέρων. Και σημαίνει ότι θα υπάρχει πιο βιώσιμη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη. Σας κατευχαριστώ για την προσέλευσή σας και θα έπρεπε να συνεχίσουμε τέτοιου είδους διαλόγους και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και σένα όλοι για τον ενδιαφέροντα αυτόν γύρο. Θα κάνω μερικά συντομότατα σχόλια. Συντομότατα. Πρώτον, τι είχαμε πει ότι θα συζητούσαμε με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο ένας ομιλητής, ο κύριος Χάνεγκαν, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πραγματική τωρινή κατάσταση της εφαρμογής του συμφώνου στις χώρες μέλη. Οι περισσότεροι όταν αναφέρθηκαν στο Fiscal Compact και τις υποχρεώσεις του μίλησαν στην πραγματικότητα για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας Ανώ το Fiscal Compact, το οποίο συζήτησε, συζητήσαμε υπό τη διεύθυνση του Ολυρέν που προσθέτει το Fiscal Compact πέραν του Συμφώνου Σταθερότητος. Το Fiscal Compact λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε τον ενωσιακό νόμο. Αυτό όμως <coughs> ισχύει ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται καμία συνθήκη που να λέει να σεβόμαστε τον ενωσιακό νόμο. Μία τροπολογία της Κομισιόν που τη δέχτηκε και το Κοινοβούλιο λέει όμως ότι ο ενωσιακός νόμος έχει προτεραιότητα επί του Fiscal Compact και μετά και το Κοινοβούλιο το δέχτηκε αυτό. Και ο Όλη Ρεν, την Προεδρία του Όλη Ρεν υπόθηκε ότι η εξισορρόπηση των προϋπολογισμών ορίζεται από τον ενωσιακό νόμο. Έχουν λοιπόν τα κράτη-μέλη την υποχρέωση να σέβονται το σύμφωνο σταθερότητας. Άρα και ευελιξία. Γι' αυτό η ευελιξία που προβλέπετε τώρα δεν έρχεται σε αντίθεση ή αντίφαση με το Fiscal Compact. Τι σημαίνει λοιπόν στην πραγματικότητα το Fiscal Compact δεν προέβλεψε τίποτα καινούριο ή διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό τουλάχιστον. Άφησε δύο κληρονομιές. Ένα είναι η ευρωδιάσκεψη και το δεύτερο η τωρινή εδώ διάσκεψη. Η τωρινή μας διάσκεψη είναι ανοιχτή και σε χώρες που δεν υπέγραψαν το Fiscal Compact όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχία. Εγώ θα βρισκόμουν σε δύσκολη θέση αν έπρεπε υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί το Fiscal Compact στο νόμο κάθε κράτους. Εντάξει, η ευρωδιάσκεψη, αυτή η διάσκεψη. Ένα απλό πράγμα λοιπόν που το είπε και όλοι Ρεν για την Τρόικα, ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η καλύτερη και η πιο αποτελεσματική. Όπως κάνει και αυτή η διάσκεψη εξάλλου. Και νομίζω καιρό είναι πια και η Τρόικα, όπως είπε όλοι Ρεν, να συμμορφωθεί με την κοινοτική μέθοδο, γιατί αυτό είναι δυνατόν, αφού δεχτήκαμε το δίμετρο, το Τούπακ και το οποίο προβλέπει λογοδοσία και έλεγχο. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι υπό άλλο πρόγραμμα και αυτό είχε προκαθοριστεί. Αλλά ήδη έχουμε εργαλεία που προβλέπουν να οργανώνονται τέτοιες συζητήσεις και αναλύσεις σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο. Σύμφωνα με τον κοινοτικό λοιπόν νόμο όπως είπαν και άλλοι, η οικονομική διαχείριση της Ευρωζώνης δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συζητήσεις σαν τη σημερινή όπως ποια θα ήταν η καλύτερη δημοσιονομική πολιτική ή φορολογική πολιτική για την Ένωση πράγμα στο οποίο δεν μπορώ μόνος μου να απαντήσω αλλά γιατί έχουμε και διαφορές απόψεων φιλοσοφικές θα έλεγα μεταξύ μας Και υπάρχουν διαφορές λοιπόν και, και μερικά δάνεια χρειάζονται, είναι απαραίτητα. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν και πρέπει να τις λύσουμε παρόλα αυτά. Αλλά η Κομισιόν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακολουθεί μία μέση οδό, προσπαθεί να συμφιλιώσει περισσότερες διορθωτικές μεταρρυθμίσεις και πιο χαλαρή λίγο δημοσιονομική πολιτική με τον σεβασμό των υποχρεώσεων εξυγίανσης μαζί όμως βέβαια με την απαραίτητη ευελιξία για να γίνει η εξυγίανση βιώσιμη ενθαρρύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως λέει και το Σύμφωνο Σταθερότητας γιατί εκεί προβλέπεται ότι οι σοβαρές μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μπορεί να εγκριθούν και με προσωρινή αποφυγή των αυστηρότερων κανόνων. Έχουμε λοιπόν διαφορές, έχουμε, έχουμε. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε και σταθερά βήματα προς τα εμπρός για καλύτερη διοργάνωση των συζητήσεων των διαφορών μας. Είναι πιο ευρωπαϊκή αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Προχωρούμε λοιπόν και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Okay, so uh, I uh, Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τη Μαρίτα Ουλστβόγκ και ε, την κυρία Άιτζα Μπάρτσα να έρθουν στην ε, Προεδρία για να ξεκινήσουμε την επόμενη συνεδρίαση που αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης.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

Dāmas Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω για τους κύκλους συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα επικοδομητικοί. Ευχαριστώ και τις και τους συναδέλφους που διήφθηναν τις πρώτες δύο συζητήσεις της σημερινής συνεδρίας. για τις επενδύσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, σε δουλειές, σε παιδεία κλπ. και στη δημοσιονομική εξυγίανση. Τώρα βέβαια ερχόμαστε στο τρίτο θέμα, η τρίτη σειρά θεμάτων, δηλαδή στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τα θέματα μας είναι σημαντικά και εξίσου σημαντικά όλα όσον αφορά την ανάγκη να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη, έχει μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη αυτή θα είναι και βιώσιμη και δεν θα αποκλεί κανένα. Έτσι μόνο θα εξασφαλιστεί ασφάλεια για το μέλλον. Η μεγάλη ύφεση που περάσαμε έδειξε ότι έλλειψη κάποιων από αυτά τα στοιχεία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και σε άτομα και σε συνολικές οικονομίες χωρών. Μπορεί ε, να σύσει μέχρι και τα θεμέλια μια κοινωνία. Αναμένεται αυτή η συμπεριληπτική ανάπτυξη, δηλαδή η μη αποκλειστική ανάπτυξη, να ενισχύσει και την πορεία της Ένωσης προς την επίτευξη των στόχων του 2020 βέβαια. Όλα τα στοιχεία, τα μακροοικονομικά στοιχεία δεν στοχεύουν στην βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη και αυτό είναι που θα μας απασχολήσει τώρα γιατί τώρα σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να περνά στην φάση της αποκατάστασης και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που, τέτοια συστήματα δηλαδή που να λειτουργούν είναι κρίσιμα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια αγορά, εξασφαλιστούν μάλλον αγορές εργασίας που να μην αποκλείουν κανένα και επίσης επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό διότι αυτού του είδους οι επενδύσεις είναι τόσο σημαντικές για τις ευρωπαϊκές χώρες για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε έναν κόσμο που αλλάζει και για να διατηρήσουν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών τους μακροπρόθεσμα. Η συμπερίληψη λοιπόν της κοινωνικής διαστάσεω σε όλους τους τομείς πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η κοινωνική συμπερίληψη είναι πολύ σημαντική. Παρόλο που η απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές εμπίπτουν βεβαίω ιδίω ε, στο πλαίσιο των εθνικών αρμοδιοτήτων και λιγότερο τη Ένωση, υπάρχει ωστόσο μεγάλο δυναμικό ανταλλαγή εμπειριών και ιδίως σε ό,τι αφορά το πώς εντάσσουν το στοιχείο της κοινωνικής συμπερίληψης οι χώρες μέλη στα μακροπροθεσμότερα σχέδιά τους. Η συμπερίληψη στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και στην ολοκλήρωση των αγορών. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να πω ότι παρότι αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για την βελτίωση του οικονομικού δυναμικού μας μέσω και μακροπρόθεσμα, βράχει πρόθεσμα ωστόσο, οι κοινωνικές τους επιπτώσεις μπορούν και είναι συχνά πολύ, μπορούν να είναι και είναι συχνά πολύ αρνητικές. Η εμπειρία της Λετωνίας έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα που οδηγούν στην ενσωμάτωση όλων παίζουν σημαντικό ρόλο για την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να εξεταστεί ποιες επενδύσεις έχουν προτεραιότητα και ποιες ενδεχόμενα να μην έχουν. Και πρέπει ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η επιρροή των επιλεκτικών δημοσιονομικών πολιτικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι και αυτό που κάνει μια χώρα μπορεί να επηρεάσει άλλες. Σε ό,τι αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις, εκεί πρέπει να αναζητήσουμε μια ισορροπία, να επιτευθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων, των υποδομών, να παρακολουθούμε όμως και την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, έτσι ώστε η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βελτιωθεί και μακροπρόθεσμα, έχοντας υπόψη βεβαίως ότι η παιδεία, οι υποδομές είναι ιδιαίτερα η παιδεία και οι υποδομές είναι σημαντικά για την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτό το κάνουμε ήδη στην Λετωνία, όπου η Βουλή μας οργανώνει συνεδριάσεις με τους Προέδρους συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών τον Φεβρουάριο και μάλιστα στις 22 και 23 Φεβρουαρίου και πληροφορούμε ότι πολλέ αντιπροσωπήσεις από διάφορε δηλώσει συμμετοχή, όχι όμω όλε. Γι' αυτό σα παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε και να έλθετε στην συνδιάσκεψη τη Ρήγα. Αξιότιμε και αξιότιμοι συνάδελφοι, ο Βάλτη Πρόσκης ακόμα δεν έχει καταφθάσει. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα δώσω τον λόγο στην πρόεδρο της ε, Επιτροπής Απασχολήσεως, κυρία Μαρίτα Ουλφσκοχ. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να κάνετε την παρέμβασή σας, αφού άλλωστε θα συμπροεδρεύσουμε στην ε, παρούσα συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένοντας τον κύριο Ντομπρόφσκης, θα επιτρέψτε μου να πω εγώ δύο λόγια για την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η οικονομική και νομισματική κρίση έφεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δοκιμασία και σε δοκιμή. 25 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και από αυτούς τα 6 εκατομμύρια είναι νέοι. 120 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να ζήσουν σε φτώχεια και σε αποκλεισμό στην Ευρώπη η συμμετοχή στην αγορά εργασίας έχει επηρεαστεί αρνητικά και η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όλα αυτά είναι πολύ μακριά βέβαια από τους στόχους του 2020, τους οποίους αποφασίσαμε πριν από λίγο καιρό. Όχι και πολλά χρόνια. Η εσωτερική αγορά με την ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αγορά και να μην οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ, σε καταχρήσεις, σε θέμα του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει δεσμευτικές προδιαγραφές για να προστατεύει τους εργαζόμενους. Ελάχιστες υποχρεωτικές προδιαγραφές, γιατί δεν πρέπει να επιδεινωθεί η κατάσταση των εργοζαμένων και να πιεστούν οι συλλογικέ συμβάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κερδίσει ποτέ, ποτέ δεν θα κερδίσουμε αν οι χώρε μέλη ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποια θα έχει τους χαμηλότερου μισθού, τους ε, εργαζόμενου με τα λιγότερα προσόντα και κακέ συνθήκε εργασία. Μια τέτοια κατάσταση εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά δεν βοηθάει επίσης και το θεμητό ανταγωνισμό. Αντίθετα, μας βάζει σε θέμητο ανταγωνισμό. Εμείς πώς θα ανταγωνιστούμε την Κίνα, τη Βραζιλία, αν έχουμε χαμηλές φιλοδοξίες όσον αφορά τα προσόντα και τις δεξιοτεχνίες των εργαζομένων. Ανταγωνισμός με χαμηλότερους μισθούς και κακές συνθήκες εργασίας οδηγούν και σε λιγότερη και χαμηλότερη αποδοχή από τους πολίτες των μέτρων αυτών. Σε αύξηση του λαϊκισμού, των εθνικισμών, στο κλείσιμο των συνόρων, πράγματα από τα οποία δεν έχει να το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό που θυμάμαι από την προεκλογική εκστρατεία πριν τις ευρωεκλογέ, το Μάιο που μας πέρασε, ήταν ένα τηλεφώνημα που πήρα από έναν ιερέα που εκπροσωπούσε την ε, Σουηδική Εκκλησία σε μια μεσαία περιφέρεια της Σουηδίας και είπε πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση λέγοντας ότι ε, σε ένα πάρκινγκ έξω από την πόλη έβλεπε πάρα πολλά φορτηγά και οδηγούς αυτοκινήτων οι οποίοι ζούσαν μέσα στα οχήματά τους. Δεν είχαν βέβαια καμία ε, συνθήκη υγιεινής, δεν είχαν θέρμανση. Η μόνη θέρμανση που είχαν ήταν από κάτι γκαζάκια που χρησιμοποιούσαν ε, για να ζεστάνουν νερό ή φαγητό. Αυτά τις παραμονές του 2015. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άλλο παρέχει πετύχει τους στόχους της. Υπάρχουν ακόμα τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών μας και η κοινωνική συνοχή βρίσκεται σε κίνδυνο εφόσον ενισχύονται οι ανισότητες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Πρέπει να ζήσουμε μέσα σε ισότητα. Είναι κομμάτι των στόχων μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην αναδιάρθρωση των κοινωνιών μας γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε ως ένωση αν δεν το πετύχουμε αυτό. Η κατανομή πλούτου, μια αξιοπρεπού ζωής, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες μας. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι όταν αυξάνονται οι ανισότητες, τότε μειώνεται και η συμμετοχή σε συνδικάτα. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι δεν μπορούν πια να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, ούτε οι συνδικαλιστές μπορούν να τους υποστηρίξουν επίσης όρις στις διάφορες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ανισότητα σημαίνει επίσης ότι μακροπρόθεσμα δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Συνεπώς όλοι έχουμε να υποφεληθούμε από ισότητα στην αγορά εργασίας, οπότε και αυτό είναι κομμάτι της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση της κρίσης και της οικονομικής διακυβέρνησης είναι κάτι που πρέπει να σέβεται την αυτονομία και την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε ήδη θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος, προς τη σωστή κατεύθυνση για την Ευρώπη. Συνεπώς, δεν πρόκειται μόνο για την οικονομία, πρόκειται και για την ισότητα, πρόκειται για την κοινωνία των πολιτών. Και ας φροντίσουμε τα πράγματα να γίνουν πιο εύκολα αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε κάτω από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Τσκόκ. Τώρα έχουμε και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τον κύριο Πιέρ Αλά Μουιέ, που ήρθε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να εναφερθούμε σήμερα στην κοινωνική διάσταση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο χαρακτήριζε τις συζητήσεις μας τις δύο μέρες που πέρασαν. Πώς να βγούμε με μόνιμο τρόπο από την ύφεση την οποία αφήσαμε να αναπτυχθεί στην καρδιά της Ευρώπης. Η πρώτη προϋπόθεση για να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομισματικής ένωσης, είναι να ενισχύσουμε και να σχεδιάζουμε μακροοικονομικές πολιτικές που διατηρούν το σύνολο των στόχων της οικονομικής πολιτικής, την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή για να αποφύγουμε αυτά τα οποία γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. 6 εκατομμύρια κόσμος έχασε τη δουλειά του. Το ΑΕΠ κάποιων χωρών μειώθηκε κατά 25% και η ανεργία των νέων έφτασε σε απαράδεκτα επίπεδα σε ορισμένες από τις χώρες μας. Η ευρωπαϊκή χρήση δείχνει ότι ο συντονισμός με δημοσιονομικούς κανόνες δεν είναι επαρκής και ότι είναι απαραίτητο στο εσωτερικό της νομισματικής ένωσης να δημιουργηθεί ένα κοινό μακροοικονομικό πλαίσιο για να προσαρμοστεί το σύνολο των πολιτικών μας στην παγκόσμια κατάσταση και στην κατάσταση στη ζώνη ευρώ. Όπως μας θύμισε ο κύριος Γιούνκερ χθε, έχουμε ανάγκη από μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης ευρώ. Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόσαμε πολιτικές λιτότητας για να ανακάμψουν τα δημοσιονομικά και να μειωθεί το κόστος της εργασίας για να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα όταν μια χώρα είναι μόνη της. Όταν όμως όλοι το κάνουν μαζί, το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή ύφεση και μια κατάσταση σχεδόν αποπληθωριστική. Όταν μια χώρα είναι μόνη της στην πρακτική μιας πολιτικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, το ηφεσιακό αν θέλετε στοιχείο ε, εν μέρει αντικαθίσταται και αντισταθμίζεται από την ανάπτυξη των εταίρων. Αλλά όταν όλοι ακολουθούν την ίδια πολιτική, τότε η ύφεση προφανώς είναι πολύ πιο σημαντική από την ανάπτυξη και το κοινωνικό κόστος είναι πραγματικά παράδεκτο στον τομέα της απασχόλησης. Μπορεί μια χώρα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του μειώνοντας το κόστος ε, της εργασίας, αλλά αυτό δημιουργεί προβλήματα στους εταίρους. Αν κάνουν το ίδιο πράγμα στην Ευρώπη όλοι, τότε δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Μια γενικότερη μείωση των τιμών, δηλαδή αποπληθωρισμός για μια ακόμη φορά. Έτσι λοιπόν χάνουμε τους στόχους, αυξάνεται η ανεργία, μειώνεται πολύ λίγο το δημόσιο έλλειμμα, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει πληθωρισμός και συνεχίζει να αυξάνεται το χρέος. 80 χρόνια μετά ξανακάνουμε δηλαδή αυτό το οποίο κάναμε στη δεκαετία του 30. Τι να πει κανεί ε, για τα ε, προβλήματα που δημιούργησε και επέβαλε η Τρόικα στην Ελλάδα. Καμία σχέση με την αλληλεγγύη που πάντα χαρακτήριζε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μπόρεσε να τραβήξει προς τα πάνω και προς την πρόοδο όλες τις χώρες που μπήκαν μέσα σε αυτήν τώρα κάνει το αντίθετο εδώ και τρία χρόνια. Όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί φοβόντουσαν, ιδιαίτερα στη χώρα μου, στη Γαλλία, ότι ο μισθολογικός ανταγωνισμός θα ε, χαμηλώσει τις αμοιβέ στις πλούσιες χώρες και θα οδηγήσει σε πολλές μετακινήσεις επιχειρήσεων. Αυτό θα συνέβαινε αν η Ευρώπη ήταν μια μεγάλη αγορά μόνο. Υπήρχαν όμως μηχανισμοί αλληλεγγύης όπως τα διαρθρωτικά ταμεία που ευνόησαν τις επενδύσεις και τον εξυγχρονισμό των νέων κρατών μελών. Έτσι λοιπόν υπήρξε μια κάποια μορφή σύγκλησης προς τα πάνω. Αν θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν μια ρύθμιση προς τα κάτω, τότε θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις πολιτικές που δεν επιτρέπουν τις συνέργειες και να ευνοήσουμε τις πολιτικές της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας που να ωφελούν τους πάντες. Πρέπει να υπάρξουν ελάχιστοι μισθοί. Ακάτα χώρα βέβαια, διαφοροποιούμενοι, για να εγγυηθούμε για την κοινωνική πρόοδο και την παραγωγικότητα να υπάρξει ένα πρώτο βασικό στάδιο κοινωνικής κάλυψης σε σχέση με την αποζημίωση για την ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης η Ευρώπη μας να ξαναγίνει ένας χώρος αλληλεγγύης και όχι μια μεγάλη αγορά η οποία θέτει σε ανταγωνισμό το ένα κράτος εις βάρος του άλλου. Η κοινωνική διάσταση των οικονομικών πολιτικών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ετήσιας εξέτασης του ρυθμού ανάπτυξης. Ένα τμήμα των συνεδριάσεων των Υπουργών Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ασχολείται με την εξέλιξη των κοινωνικών πραγμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα κοινωνικό Eurogroup, το οποίο θα μπορεί να κάνει συστάσεις και για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε στη ζώνη ευρώ. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι σήμερα γιατί η Ευρώπη βάζει την απασχόληση και την ανάπτυξη στο κέντρο των στόχων της. Η Κεντρική Τράπεζα προχωρά με το δικό της πρόγραμμα νομισματικής διευκόλυνσης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά το σχέδιο αυτό 315 δις σε τρία χρόνια. Ε, Φιλόδοξο ακούγεται βέβαια λόγω της υπερβολικής μόχλευσης, αλλά παρόλα αυτά σε σχέση με τις ανάγκες δεν είναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εξωτερικό πλεόνασμα 230 δις που δεν οφείλεται στην ανταγωνιστικότητα, αλλά στην πτώση της εσωτερικής ζήτησης. Αυτή η αποτεμίευση των 230 δις κατέτος δείχνει ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης χωρίς πρόβλημα χρηματοδότησης. Η εσωτερική αποταμίευση στην Ευρώπη θα το καλύψει. Πρέπει η Ευρώπη λοιπόν να ξαναβρει τη στρατηγική της Λισαβόνας και το πνεύμα της, βάζοντας στο εσωτερικό της οικονομικής της πολιτική τους πέντε στόχους της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Απασχόληση, έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση, μείωση της φτώχειας και καταπολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Και μιας και χαράξαμε σε πέτρα, σε μάρμαρο, τους κανόνες και τα κριτήρια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να κάνουμε και το ίδιο πράγμα για τα κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν την ίδια ισχύ με τα πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα. Αυτό το θύμισε πριν λίγο καιρό ο Ματέο Ρέντσι, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ακόμα και η προγραμματική δήλωση του γερμανικού συνασπισμού το ίδιο έλεγε θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ισότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Να είναι στο ίδιο επίπεδο με την ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Όμως συνάδελφοι, οι μεμονωμένοι εγωισμοί και οι ανισότητες οδήγησαν στα προβλήματα της κρίσης του 2008. Η έλλειψη αλληλεγγύης ανάμεσα στα έθνη είναι εν μέρη υπεύθυνη για το μέγεθος της κρίσης στη ζώνη ευρώ. Βάζοντας ξανά λοιπόν την αλληλεγγύη στην καρδιά της νομισματικής μας ένωσης θα μπορούμε μόνιμα να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντομπρόφσκι, στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινωνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρία Ουλσκοκ, κύριε Μέ, κύριε Γκί Ράιντερ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κυρίες και κύριοι, Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να συμμετάσχω και εγώ στην κοινοβουλευτική αυτή εβδομάδα και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Έχει μεγάλη σημασία διότι η κοινοβουλευτική αυτή εβδομάδα καταδεικνύει το κοινό μας ενδιαφέρον να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση όχι μόνο μέσα στην Ευρωζώνη αλλά σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα συζητήσατε ήδη τους τρεις πυλώνες των νέων οικονομικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως διατυπώθηκαν στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης του 2015. Ενίσχυση των επενδύσεων μέσω του επενδυτικού πακέτου 315 δισεκατομμυρίων του κ. Γιούγκερ, νέα δέσμευση υπέρ διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Αυτοί οι τρεις πυλώνες θα μας βοηθήσουν να βάλουμε και πάλι στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη και να της προσφέρουμε νέες θέσεις απασχόλησης και ανταγωνιστικότητα. Σήμερα μας δίνεται ευκαιρία να συζητήσουμε το τι θέλουμε να πετύχουμε με τους τρεις αυτούς πυλώνες. Την, ε, τις κοινωνικές αγορές, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Από την κρίση και μετά, από το 2008-2009 δηλαδή, κοινωνικές αποκλίσεις έγιναν ακόμα μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Το ποσοστό ένδυας, ανεργίας, ιδίως των νέων, αυξήθηκε και το χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί κατά πολύ. Αυτό βέβαια υπονομεύει τους ίδιους τους στόχους του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος που είναι η σύγκληση και βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλους τους Ευρωπαίους. Αγορές εργασίας που δυσλειτουργούν, φτωχή κοινωνική δίκτυ σε μία χώρα μέλος είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί όλες τις χώρες μέλη. Διότι υπάρχουν επιπτώσεις διασυνοριακές στις γείτονες χώρες και ακόμα παραπέρα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνδυάζοντας την ανάπτυξη δεξιοτεχνών προσόντων με την αγορά απασχόλησης. Κατά τη γνώμη μας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι μόνο οικονομική, έχει μεγάλη σημασία απασχόληση, οι κοινωνικοί δείκτες. Αλλιώς δεν γίνεται. Οι απασχόληση κοινωνικές πολιτικές έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και το ένα ενισχύει το άλλο. Για να λειτουργήσει καλά η ΟΝΕ, οι διευθυντικές της δομές πρέπει να συμπληρωθούν για να πάψουν να υπάρχουν οι τελευταίες διαφορές που υπάρχουν και να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε με τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί, να τα προσαρμόσουμε και να φροντίσουμε να είναι αποτελεσματικά. Έχει ήδη γίνει αρκετή δουλειά. όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση του 2013 για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Θα αναφέρω σε διάφορα στοιχεία. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε ότι η απασχόληση και η κοινωνική διάσταση πρέπει να παίζει μεγαλύτερο ρόλο σε ένα γενικότερο και μακροπρόθεσμο ε, σχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης αγάγαμε και τον πίνακα επιδόσεων όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες και την απασχόληση, ακριβώς για να ενισχυθεί ο συντονισμός της απασχόλησης με τις κοινωνικές πολιτικές μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Συγχρόνως προσθέθηκαν και διάφοροι συμπληρωματικοί κοινωνικοί δείκτες. Τα βήματα που διαθέτουν οι κοινωνικοί εταίροι για διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιούνται περισσότερο ώστε να εμπλακούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την τριμερή διάσκεψη κορυφή και τον οικονομικό και κοινωνικό διάλογο. Υπάρχουν και διάφορες προτάσεις που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2015. Ενίσχυση της απασχόλησης σε σχέση με την ΟΝΕ. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο στο πακέτο της ΟΝΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση στο Συμβούλιο του Ιουνίου με προτάσεις. Δεύτερον, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Να μην υπάρχουν καταχρήσεις και αυτό θα γίνει συντονίζοντας ακόμα καλύτερα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Τρίτον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει πακέτο για περισσότερη ολοκλήρωση και διασημότητα της αγοράς εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν περισσότερες δεξιοτεχνίες και προσόντα. Στη συνέχεια, συμμετοχή των ε, εθνικών κοινοβουλίων. Πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας για να είναι πιο ε, κυκλικά και αυτό πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Να ενισχυθούν οι προσλήψεις. Να προστατεύσουμε το κοινωνικό μοντέλο με αποτελεσματικότερα συστήματα, να αποφύγουμε τους κινδύνους, να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και τα προσόντα των πολιτών, οι οποίοι θα έχουν διαβίου κατάρτιση, ώστε να προσαρμόζονται στις αγορές εργασίας. Θέλουμε ενίσχυση λοιπόν της απασχόλησης και ανάπτυξη ενισχύοντας και προσφέροντας κίνητρα για νέες, για δημιουργία δηλαδή θέσεων απασχόλησης. Πέρα από τις προτάσεις που σας περιέγραψα μόλις τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και πιο μακροχρόνιες φιλοδοξίες στον κοινωνικό τομέα. Για να είναι βιώσιμη η ΟΝΕ πρέπει να πετύχει μεγαλύτερη σύγκληση. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι ευκαιρίες μας προσφέρει ο ετήσιος κύκλος οικονομικών, οικονομικού συντονισμού που είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η ΟΝΕ πρέπει να διασφαλίσει την συμμετοχή όλων. Να μην υπάρχουν αποκλεισμοί Θέλουμε να μειωθεί η ένδια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επίσης την ανεργία με μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση που να περιλαμβάνει επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, στη δημιουργία ενός ε, επιχειρηματικού πλαισίου που να είναι ευνοϊκό για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο από τον κοινωνικό διάλογο και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις χώρες μέλη. Όταν ήμουν στην ε, Λετωνία είδα και εγώ πόσο ανάγκη έχουμε για κοινωνικό διάλογο και πόσο ο παράγοντας αυτός, ο κοινωνικός ε, διάλογος δηλαδή, βοήθησε τη Λετωνία να βγει από την οικονομική κρίση είναι απόλυτα θεμητός και δημοκρατικός τρόπος για να έχουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη οι δράσεις μας. Όπως έχω ξαναπεί εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο και προκειμένου η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ενισχυθεί περισσότερο στο τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Προβλέπουμε μια διάσκεψη κορυφής με τους κοινωνικούς εταίρους μας της Μαρτίου φέτος και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε εκεί τις σχέσεις μας με τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουμε εκφράσει τις ε, απόψεις μας Όσον αφορά τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους, έχουμε πει ότι πρέπει να συμμετέχουν ακόμα περισσότερο. Και αυτή η κοινοβουλευτική εβδομάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ένας τέτοιος ισχυρός διάλογος πρέπει να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση και να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις και σχόλια έχετε. Σας ευχαριστώ και τον Μπρόφσκης. Ο επόμενος ομιλητής στη συνεδρία αυτή, ο Γενικός Διευθυντής του ILO. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εσείς συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να συνομιλήσω μαζί σας στη σημερινή συνάντηση που είναι και επίκαιρη και καλή ευκαιρία διότι πιστεύω ότι οι προκείμενες περιστάσεις είναι επίγουσες για την ενίσχυση της κοινωνικής διαστάσεως της ε, Οικονομικής και νομιματικής Ενώσεως και ελπίζω ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας να μπορέσει να συμβάλλει. Η ενίσχυση της ε, Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να παραγάγει προϊόν προς όφελος όλων. Και αυτό έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Βελτίωση δηλαδή του βιωτικού επίπεδου και κάποιο βαθμό σύγκλησης. Έτσι λοιπόν μεταξύ 1999 και 2007 η μέση ανεργία στις 12 αρχικές χώρες μειώθηκε κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες και οι διαφορές στους καλύτερους και στους χειρότερους μαθητές της τάξης ήταν περίπου της τάξης του 5,5%. Αυτή ήταν η εποχή όπου πραγματικά πρόσφερε κοινή ευημερία ε, η Οικονομική Ένωση. Όμως η κρίση που άρχισε το 2008 αντέστρεψε τις τάσεις αυτές. Αυξήθηκε η ανεργία και μάλιστα απότομα και πάνω από τα όρια που ίσχυαν στην ε, Ένωση πριν. Και τώρα οι διαφορές είναι της τάξης του 22% μεταξύ των χειρότερων και των καλύτερων. Η σύγκληση λοιπόν υποχώρησε έχει παραχωρήσει τη θέση της σε βαθιές ανισότητες και η κοινή ευημερία έχει αντικατασταθεί από ευρεία πόλωση και αποκλεισμό. Άρα δεν είναι εκπληκτικό ότι έχει υποσκάψει πλέον την υποστήριξη του κόσμου για την οικονομική και νομισματική ένωση ΟΝΕ. Και οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάει το ερώτημα δεν είναι αν θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, αλλά πώς. Και αν τα πράγματα έχουν έτσι, θα πρέπει νομίζω να λάβουμε δράση σε δύο επίπεδα. Πρώτο, να ενισχύσουμε τα μέτρα στο επίπεδο των χωρών για τις ε, αγορές εργασίας με τρεις προτεραιότητες. Πρώτο, να ενισχύσουμε την μετάβαση από το σχολείο στο επάγγελμα. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την υποστήριξη σε αυτούς που ζητούν εργασία και ιδίως τους μακρόχρονα άνεργους. Τρίτο, να υποστηρίξουμε την διατήρηση της απασχόλησης σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοκ απ' έξω. Πολλά παραδείγματα για ε, εθνικές επιτυχίες υπάρχουν σε ορισμένους από τους τομείς αυτούς. Η προσοχή στην ποιότητα της απασχόλησης θα κάνει την ευρωπαϊκή οικονομία και πιο ανθεκτική και πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Έτσι λοιπόν η αύξηση της ε, παραγωγικότητας και σε, ε, σε όλες τις χώρες θα πρέπει να είναι ε, ένας στόχος. Η εξελίξη που είδαμε και στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, η προστασία των ευάλωτων θέσεων εργασίας όπως στην Ισπανία, η διευκόλυνση ε, εξέβρεση εργασίας σε σταθερές ε, απασχολήσει όπως στην Αυστρία. Η θέσπιση κατώτατων εισοδημάτων στα ανάλογα επίπεδα με την εμπλοκή των εργοδοτών έχουν όλα οδηγήσει σε επιτυχίες στην Ευρώπη όπου άρχισαν να εφαρμόζονται και ήδη τα μιμούνται και με αρκετή επιτυχία και εκτεταμένα μάλιστα άλλες περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα Όλα αυτά βέβαια έχουν κρίσιμη σημασία. Αλλά ακόμα και ενισχυμένες προσπάθειες των ίδιων των χωρών δεν θα αρκίσουν από μόνες τους. Μία αποτελεσματική κοινωνική διάσταση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο συνολικής προσέγγισης της ΟΝΕ που θα βασιστεί στα ήδη φυστάμενα μέτρα και σε εποπτικούς μηχανισμούς. Χρειάζεται να αντιμετωπιστούν καλύτερα καταστάσεις ασύμετρων σοκ, ασύμετρων κραδασμών που θίγουν ορισμένες χώρες, τις πλήττουν δηλαδή περισσότερο από άλλες. και όπου οι χώρες της ΩΝΕ που δεν μπορούν να υποτιμήσουν το νόμισμά τους αναγκάζονται να προχωρούν σε εσωτερική υποτίμηση μειώνοντας τους μισθούς, τις συντάξεις και βεβαίως υπονομεύοντας και τη σταθερότητα της ίδιας της ΩΝΕ το σημείο αφετηρίας θα μπορούσε να είναι η χρήση των υφιστάμενων θεσμών, όπως των διαρθρωτικών ταμείων και της εγγύησης των νέων, για να στοχεύσουμε σε μια προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων. Να αναβαθμιστούν τα μέτρα αυτά, ώστε να παρακολουθούν την, τις διακυμάνσεις της πορείας της απασχόλησης. Ορισμένοι μάλιστα είπαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν να γίνουν και μηχανισμοί ανακατανομής βεβαίως με την απαραίτητη αιρεσιμότητα. Πρέπει να στοχεύσει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δουλειές ε, και εντιμότητα και αυτό είναι μια εγγύηση ήδη και στο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων που ανακοίνωσε η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα από τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθεί. Ο ΆΕΛΟ εξέτασε το δυναμικό Δημιουργία απασχόλησης του σχεδίου επενδύσεων τη Επιτροπή Γιούνκερ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν βασιστεί στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εάν ληφθούν υπόψη τα εφιστάμενα επίπεδα ανεργίας, εάν οι επενδύσεις βελτιωθούν, τότε το σχέδιο μπορεί εν τέλει να οδηγήσει στη δημιουργία 2,1 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης μειώνοντας έτσι το, τη συνολική ανεργία στην Ευρώπη κατά μια ποσοστία μονάδα. Αυτά όμως θα αποδώσουν, αλλά δεν είναι και αναπόφευκτα έτσι. Εξαρτάται από, το εάν θα συμπεριληφθεί η κοινωνική διάσταση στο σχέδιο επενδύσεων. Από αυτές τις πρωτοβουλίες προκύπτουν πολλά θέματα και πολλά άλλα θα μπορούσαν να προσθεθούν σε αυτά. Ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας και απασχολήσεως μπορούν να μπουν και μέσα στις εποπτικές διαδικασίες της ΟΝΕ με στόχο να υπάρξει μια ανταγωνιστική ΟΝΕ και επίσης οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν έτσι ώστε να δώσουν νέα όθηση στον κοινωνικό διάλογο μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ασφαλώς το σωστό μείγμα πολιτικών και οι σωστές διαστάσεις τους παίζουν μεγάλο ρόλο για τους δημοκρατικούς θεσμούς και οφείλουν σε αυτούς να συζητηθούν και από αυτούς να εγκριθούν. Τελειώνοντας, έχω ένα μήνυμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο. Ήδη συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη, ιδίως αυτές που θίγονται περισσότερο από την ανεργία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδουμε μεγάλη αξία στις συνεργασίες αυτές και νομίζουμε ότι μπορούν να αποδώσουν ιδίω λόγω των αξιών που συμμεριζόμαστε. Ο ILO θα ενισχύσει τον, διάλογο, τον κοινωνικό διάλογο όπου θεωρεί ότι αυτός έχει μειωθεί με επιθεωρήσεις εργασίας, με τον αγώνα κατά της αδίλωτης εργασίας, με την προστασία των συστημάτων ε, κοινωνικών ασφαλίσεων και όπου αλλού χρειάζεται διότι η ΟΝΕ προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας και ελπίζω θα μπορέσουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσατε τους ομιλητές μας. Τώρα λοιπόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάπως σύντομα τη διαδικασία για να πάρετε το λόγο. Πολλούς έχω ήδη στον κατάλογο μιλητών από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως και σήμερα το πρωί και νωρίτερα. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Δύο λεπτά το πολύ ο καθένας. Αν υπάρχουν κι άλλοι που θέλουν το λόγο, τότε έχετε μπροστά σας τις κάρτες με τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε το λόγο, συμπληρώστε τις και δώστε τις σε κάποιον κλητήρα. Εκπρόσωπος του Σλοβενικού Κοινοβουλίου πρώτο, κύριο Πράνκα. Παρακαλώ. Σποστοβάνε, Spoštovana Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ. Καταρχήν, καταρχήν λέγω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση αυτής της διάσκεψης. Την κοινωνική διάσταση Ίσως θα έπρεπε να την είχαμε συζητήσει στην αρχή και όχι στο τέλος της εκδήλωσης, γιατί έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για μένα και για αντικειμενικούς λόγους. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος τόσο και λιγότεροι είναι παρόντες. Παρ' όλα αυτά οι διήμερες συζητήσεις μας έδειξαν τη σημασία που έχει, τη σημασία λέγω που έχει το θέμα. Τελεία. Είναι τώρα σαφές τι Ευρώπη θέλουμε η σημασία του λεγόμενου τριγώνου, δηλαδή προϋπολογισμούς, επενδύσεις κλπ. Σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ακόμα μια διάσταση, την τέταρτη. Απασχόληση και κοινωνικές ασφαλίσεις. Πρέπει να τονίσουμε την κοινωνική ασφάλιση. Πρώτον, ε, προσωπικά, θα ήθελα να υπάρξει περισσότερη κοινωνική ασφάλεια και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνούσαν και πολλοί άλλοι. Παρά τις πολιτικές μας διαφορές. Νομίζω ότι η λύση στο πρόβλημα αυτό έγκυται στη δημιουργία θέσεων υψηλής ποιότητας. Δεν είμαι κατά και της ευελιξίας ή της λεγόμενης ασφαλιξίας, γιατί μπορεί και αυτό να προσφέρει ορισμένες δυνατότητες για μεγαλύτερη ασφάλεια εκείνων που ήδη έχουν απασχόληση. Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάτι. Για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η διασύνδεση διαφόρων πολιτικών. Την πολιτική απασχόλησης με την πολιτική παιδείας, στέγασης και άλλων. Επιτρέψτε μου κύριοι συνάδελφοι να καταλήξω με τα ακόλουθα λόγια. Τα κατώτατα πρότυπα για την απασχόληση δεν αρκούν. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για τα βέλτιστα πρότυπα και όρια. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει πολυπολιτιστική και κοινωνικά δίκαια ένωση για όλους τους πολίτες. Γιατί κάθε αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο αδύνα, πιο αδύνατος της κρίκος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, επόμενος ομιλητής, ο εκπρόσωπος της Λιθουανίας, ο κύριος Φατσαρίντικος. Και μετά, ο εκπρόσωπος της Γερμανίας, ο κύριος Χούμπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητούμε το τελευταίο μας θέμα της κοινοβουλευτικής αυτής εβδομάδας που είναι, έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Εχθές και σήμερα το πρωί μίλησαμε για άλλα θέματα και αυτό το έχουμε βάλει τελευταίο. Ελπίζω όμως ότι θα γίνει το πρώτο στο μέλλον. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Δύο πτυχές θέλω να συζητήσω του θέματος. Πρώτον, το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων και δεύτερον η ανέχεια. Είχαμε πει ότι η κινητικότητα είναι από τις κύριες αξίες της ευρωπαϊκής άνεσης, αλλά να ισχύει για όλους. Για όλους. Η νομισματική ένωση και η ενδυνάμωση της κοινωνικής της διάστασης δεν μπορούν να παραμείνουν προτεραιότητα εάν πολλοί άνθρωποι όπως οι συμπολίτε μου εμποδίζονται από την κοινωνική τους κατάσταση. Είναι άνθρωποι που η χώρα έχει εκπαιδεύσει αλλά αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους για να πάνε σε άλλες χώρες μέλη της Ένωσης διότι υπάρχει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Η διαφορά μεταξύ του πλούτου είναι τεράστια. Αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε σε άλλες χώρες μέλη δημιουργούν πλούτο σε αυτές τις άλλες χώρες μέλη. Και αν και οι μετανάστες υπάρχουν, τη χάνουν κακής μεταχείρισης και τους ψέγουν για τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας από τους λαϊκιστάς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι προσβολή και για εκείνους και για τις κοινέ αξίες της Ένωσης. Και τώρα για την ανέχεια. Δεν θα ήθελα να τη συζητήσω λεπτομεριακά γιατί μόνο ένα πράγμα θέλω να τονίσω. Το όριο της ανέχειας σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Ας πούμε οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία στη Σουηδία είναι πολύ ψηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα και τη Λιθουανία που είναι ακόμα χαμηλότερη και οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν αντίστοιχο ύψος και διαφορές. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα κοινωνικής ασφάλειας σε κάθε χώρα μέλος και σε ενωσιακό επίπεδο. Επομένως, η σημαντικότερη προτεραιότητα για μας είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης σε όλες τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοώ καλά ότι όλοι όσοι συμμετέχετε στη συζήτηση θεωρείτε τα διάφορα κοινωνικά θέματα ως πολύ σημαντικά βεβαίως, αλλά θα σας παρακαλέσω όλες και όλους να τηρείτε τα χρονικά όρια των παρεμβάσεων. Άλλωστε αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε όλες και όλοι τις τελευταίες αυτές δύο ημέρες. Διότι έχουμε πάρα πολλούς διαγραμμένους ακόμη. Από τη Γερμανική Βουλή ο κύριος Χόμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μιλούμε για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό νομίζω είναι απαραίτητο και κατεπήγον. Και συμφωνώ με τους δύο προλαλήσαντες, θεωρώ ότι η ενίσχυση της διάστασης αυτής πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Εάν αναλύσουμε το status quo, που βρισκόμαστε σήμερα στην ΟΝΕ, διαπιστώνουμε ότι εφαρμόζονται διάφορα κριτήρια στην αξιολόγηση. Έχουμε τα δημοσιονομικά κριτήρια Μερικοί λένε, α, κοιτάξτε, έχουμε κάποια πρωτογενή πλεονάσματα, αρχίζουμε να βγαίνουμε από την κρίση. Αν τα εξετάσουμε όμως από άψη κοινωνικής πολιτικής, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Βρισκόμαστε ακόμα στα όρια της ύφεση, βρισκόμαστε μπροστά σε, μια, σε έναν αποπληθωρισμό, ευχαριστώ και τον Γάλλο συνάδελφο που το τόνισε αυτό προηγουμένως, Άρα, ήδη τα πράγματα είναι πολύ εύθραυστα από αυτή την, από αυτή την άποψη. Αν εξετάσουμε τώρα την κοινωνική διάσταση, εγώ θα πω ότι βρισκόμαστε σε καταστροφική κατάσταση. Σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, αυτό ελέγχθη κατ' επανάληψη, και ευχαριστώ ε, ήδη εκείνες και εκείνους που το τόνισαν, η ανεργία των νέων στην Ισπανία, στην Ελλάδα, είναι τη τάξη του 50% και σε άλλες χώρες όπως Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρο, άνω του 30% και ούτω καθεξής. Η ιδέα ανεργία στο σύνολό της είναι υψηλότερη από ό,τι στην αρχή της ΟΝΕ. Αυτό αποτελεί πραγματικό σοκ αν το σκεφτεί κανείς. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κατεπηγόντως να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση. Με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θεσπίσαμε με νομοθετικό τρόπο εργαλεία τα οποία στοχεύουν άμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία. Έχουμε όμως πολύ αδύναμα εργαλεία εντό εισαγωγικών για τον συντονισμό μιας οικονομικής πολιτικής αντιμετώπιση των ελλημάτων κλπ. Και πάρα πολύ αδύναμους μηχανισμούς σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση. Υπάρχει το λεγόμενο βαθμολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ακούστηκε που είναι πιο πολύ το θερμόμετρο με το οποίο μετρούμε την θερμοκρασία του ασθενούς αλλά δεν μας επιτρέπει να κάνουμε διάγνωση ούτε θεραπεία, ούτε είναι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας. Υπάρχουν και κάποια προγράμματα τα οποία υποστηρίζω και εγώ, όπως το πρόγραμμα εγγύησης για τους νέους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματικά δραματική στροφή και ιδίως η εξελίξη των τελευταίων ημερών και στην Ισπανία και στην Ελλάδα δείχνουν προς τα που πρέπει να πορευτούμε. Θα ρωτήσω τον κύριο Ράιτερ από τον πρόεδρο του ΑΕΛΟ πώς κρίνει την κατάσταση στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, το δικαίωμα σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Γνωρίζω ότι ο ΑΕΛΟ δραστηριοποιήθηκε εκεί, στον τομέα αυτό και στη χώρα αυτή πρόσφατα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σα, λέει η και θα ακολουθήσει η Ευρωβουλευτής κυρία Ροδρίγες, την οποία θα ακολουθήσει ο εκπρόσωπος της Εστονικής Βουλής, κύριος Κάλεμπετ. Σας ευχαριστώ για την ποιότητα του πάνελ. Η Νομισματική Ένωση είναι ο κινητήρας αλλά δυστυχώς δεν ασχολείται ο κινητήρας αυτός με το να θέσει σε κίνηση την κοινωνική Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα απασχόληση σε ορισμένες χώρες, άλλες έχουν προβλήματα με το κοινωνικό ντάμπινγκ και αυτά είναι οι δύο πλευρέ του ιδίου νομίσματος βέβαια. Απαιτείται εμεί να εφαρμόσουμε καλύτερα κοινωνικά επίπεδα προστασίας, σωστές και δραστήριε κοινωνικέ πολιτικέ. Και αυτό δεν αρκεί καν. Πρέπει να πάμε στην πηγή του προβλήματος. Έτσι ώστε να, επιτρέψουμε σε όλες τις χώρες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην πίστοση και να μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας και να ανοίξουν τη χώρα αυτούς για επενδύσεις. Στα πλαίσια της Ένωσής μας απαιτείται ένα αποτελεσματικό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει βέβαια και την αντίστοιχη και κατάλληλη δημοσιονομική ισχύ. Έτσι θα καταστήσουμε τις πολιτικές μας ικανές να προχωρήσουν και να εφαρμοστούν σύμφωνα πάντα και με τα κέρδη σε επίπεδο παραγωγικότητας. Όλα κρίνονται από την κοινωνική διάσταση της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι Στη φάση αυτή θα ζητήσουμε από τους βασικούς ομιλητές να δώσουν κάποιες πρώτες απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι η ανεργία ποικίλει από 4,8% στη Γερμανία σε 25,8% στην Ελλάδα. Η ανεργία είναι το πιο σημαντικό, αν θέλετε, κοινωνικό στοιχείο. Και για την Ευρώπη, έτσι ώστε να φροντίσει η Ευρώπη να βρει θέσεις απασχόλησης στους πολίτες της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει ευτυχής για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η ευρωπαϊκή πολιτική οι στόχοι για την Ευρώπη του 2020 δεν συνδέονται δυστυχώς τόσο στενά όσο θα έπρεπε με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για υψηλότερα επίπεδα ανακατανομής σε διάφορες χώρες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να δούμε αν κάτι τέτοιο μπορεί να είναι παραγωγικό ή όχι. Η υπερβολική ανακατανομή πολλές φορές καταστέλει την επιχειρηματικότητα και εμποδίζει την ανάπτυξη με ικανούς ρυθμούς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν δημιουργεί το κράτος τις θέσεις. Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν και τον δημόσιο τομέα και προσφέρουν αξία τη θέμενη βελτιώνοντας τις κοινωνικές συνθήκες. Σας ευχαριστώ κύριε Κάλμετ. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ντομπρόφσκης. Έχουν τεθεί αρκετές και σοβαρές ερωτήσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα δώσετε τις απαιτούμενες απαντήσεις. Πράγματι, συνάδελφοι, τέθηκαν αρκετές σημαντικές ερωτήσεις. Και κάποιες από αυτές θα προσπαθήσω να απαντήσω. Έγιναν ερωτήσεις σχετικά με το στοχολόγιο κοινωνικών δικτών και πώς λαμβάνουμε υπόψη μας αυτές τις κοινωνικές πληροφορίες στο σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Να πω εδώ ότι με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο οι δείκτες αυτοί λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και εννοώ τους κοινωνικούς δείκτες ιδιαίτερα όταν προετοιμάζουμε τις ε, ειδικέ ανακράτως στάσεις υπογραμμίζουμε τις ανισότητες οι οποίες μπορεί να ισχύουν σε ορισμένες χώρες. Στόχος των δικτών αυτών είναι να ισορροπήσουμε καλύτερα τις οικονομικές πολιτικές από τη μία με τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης από την άλλη. Βεβαίως, απαιτείται να ενισχύσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Έτσι μόνο θα βρεθεί λύση στα προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανεργία είναι ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει όμως να το δούμε αυτό όχι μόνο με βάση τους οικονομικούς δείκτες αλλά και μέσω της λεγόμενης κοινωνικής στήριξης για την επίτευξη κάποιων ε, στόχων στον κοινωνικό τομέα. Σήμερα η Επιτροπή ε, πρότεινε την αύξηση των πιστώσεων για την εγγύηση για τους νέους αυτό είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει 20 χώρες που είναι επιλέξιμες ε, για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Χώρες ε, στις οποίες ε, η ανεργία των νέων είναι άνω του 20-25% σε μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Με την πρότασή της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει περίπου ένα δις κατά τη διάρκεια του 2015 στα πλαίσια της χρηματοδότησης του, αυτού, του μέσου. Ελπίζουμε η πρόταση αυτή να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και με τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά μέσα. Αυτό το είπα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Είπα επίσης ότι όταν συζητάμε το θέμα της εμβάθυνσης της Οικονομικής Ένωσης, ένας από τους βασικούς στόχους θα πρέπει να είναι η σύγκληση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική σύγκληση. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μια διαρκής λύση στο πρόβλημα της κρίσης. Σε ευχαριστούμε κύριε Ντομπρόσκης. οι συνάδελφοι από τη Σλοβενία, Εσθονία, Γερμανία και άλλοι έκαναν σχόλια τα σχόλιά τους και τώρα ο εκπρόσωπος του ΙΕΛΟ. Έχετε τίποτε να προσθέσετε ή να απαντήσετε σε κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε με ρώτησαν, μου ρώτησαν κάτι πολύ συγκεκριμένο για την Ελλάδα. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας έχει δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω δύο-τρία σχόλια για την εμπειρία μας ως προς αυτήν την εμπλοκή του. Ένα από τα πιο ατυχή στοιχεία της ελληνικής μας εμπειρίας ήταν ότι ο κοινωνικός διάλογος στη χώρα αυτή έχει σταματήσει απλώς δεν έχει περάσει το stress test θα έλεγα της ε, συνεννόησης των κοινωνικών εταίρων και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να παίξουν το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν παρά ή λόγω των ε, παρεμβάσεων της Τρόικας. <clears throat> Τι είδαμε στην Ελλάδα. Τελείως καινούργιες μορφές εργασιακών σχέσεων σχεδόν καταστροφή των συλλογικών συμβάσεων, αλλά αυτό δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη μείωση των μισθών και για μας είναι σημαντικό να τα ξαναδούμε όλα αυτά, γιατί κάναμε προσπάθειες να επανέλθουμε στον κοινωνικό διάλογο. Έγινε μια συνάντηση στη Γενέβη του τότε Υπουργού Εργασίας, με τον τότε Υπουργό Εργασίας και καταλήξαμε <coughs> σε, συμφωνία για ορισμένα θέματα όπως τις διαδικασίες για τις συλλογικές απολύσεις που είναι πολύ σημαντικό θέμα στην Ελλάδα. Ό,τι και να θεωρεί κανείς για το περιεχόμενο της συμφωνίας, το ότι έγινε εκείνος ο διάλογος ε, είναι σημαντικό για το μέλλον. Σαφώς χρειάζεται να γίνουν περισσότερα ως προς την Ελλάδα. Ίσως να επαναλάβω αυτά που είπαν κι άλλοι όσο έχω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος δηλαδή, είναι πολύ σημαντική η σύγκληση. Η νομισματική ένωση πρέπει να δημιουργήσει σύγκληση για όλα τις τα μέλη και θα ήθελα επίσης να τονίσω αυτά που υπόθηκαν για την μεταχείριση των ξένων εργαζομένων, των μεταναστών πρέπει να είναι ίση και δίκαια αυτή η μεταχείριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για την κοινωνική ασφάλεια και την ανάγκη ίσης μεταχείρισης ως προς αυτό στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων θα έχει κάτι να μας πει. Και γι' αυτό δίνω το λόγο, της δίνω το λόγο. Πώς σχολιάζεται αυτό το θέμα και τα ερωτήματα από τους πέντε ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να μιλήσω για το ότι την κοινωνική διάσταση την συζητήσαμε και την πρώτη μέρα και την πρώτη διότι πρέπει φυσικά να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτά τα θέματα εγώ είμαι προεδρεύουσα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων εδώ στο Κοινοβούλιο και για μας είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ως προς αυτό σύγκληση. Παραδείγματος χάρη πρέπει να είμαστε σαφέστατοι ως προς το ότι μιλάμε για ίσους μισθούς, για ανάλογες συνθήκες στους εργαζόμενους. Ανεξάρτητα από το από πού προέρχεται ο εργαζόμενος. Αν κανείς είναι από τη Σουηδία και εργάζεται στην Πολωνία ή το αντίθετο αν είναι από την Πολωνία και εργάζεται στη Σουηδία πρέπει να ισχύουν τα ίδια για ανάλογες συνθήκες. Το θέμα είναι η εργασία που εκτελείται και όχι το από πού προέρχεστε. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αναγνωρισμένη αρχή αλλά δεν εφαρμόζεται 100%. Είναι όμως σημαντικό να μην δημιουργηθεί μισθολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών. Διότι για ίση εργασία πρέπει να υπάρχει ίση ίσως μισθός. Det är Για την ακτοπλοεία. Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιηθεί η ακτοπλοεία, αλλά δεν δουλεύει, δεν έχει αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε φοβερή κατάχρηση και παραβίαση των κομμάτων των εργαζομένων. Βλέπουμε και εγκληματική δραστηριότητα, βλέπουμε θέματα ασφαλείας στις μεταφορές, βλέπουμε σαφέστατα ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ οδηγών, εταιριών, μεταφορών κτλ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι κανόνες για την ακτοπλοϊκή μεταφορά πρέπει να εφαρμόζονται με το πνεύμα για το οποίο είχαν γραφτεί. Αλλιώς θα υπάρχουν όλο και περισσότερα προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα μάλιστα, μεταξύ των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Ακόμη λοιπόν πρέπει να γίνουν πολλά για την κοινωνική διάσταση. Το θέμα είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες εργασίας ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Αυτό θα το ξαναδούμε βέβαια σε αυτή τη θητεία και δεν πρέπει να επιτρέψουμε την κρίση που βλέπουμε μπροστά μας να υπονομεύσει αυτά τα βασικά δικαιώματα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και όλοι μας ή οι περισσότεροι από μας εργάζονται, είναι εργαζόμενοι δηλαδή και απασχολούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχουν το, ίσο, το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων και αξιοπρεπίας από όπου και αν προέρχονται. Αυτή πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή μας εδώ στο Κοινοβούλιο και ξέρω ότι πάρα πολλοί βουλευτές από πολλές χώρες το υποστηρίζουν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος. Ο κύριος Λεμουέ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε Λεμουέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι όσοι πήραν το λόγο σήμερα υπογράμμισαν πολύ σωστά την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη. Είναι και η ιστορία των ευρωπαϊκών εθνών. Ποτέ δεν κάναμε διάκριση του ενός από το άλλο. Αυτό που πάντα χαρακτήριζε την Ευρώπη είναι ακριβώς το κοινωνικό της μοντέλο ή τα κοινωνικά της μοντέλα, γιατί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, που εξελίχθηκαν σιγά σιγά συγχρόνως με την οικονομική ανάπτυξη. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα το κατάφερε επίσης αυτό. Να τα συνδέσει δηλαδή παρόλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο με την παγκοσμιοποίηση που συχνά μεγαλώνει τις διαφορές μεταξύ των χωρών, παρόλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν οι διαφορές αυτές ανάμεσα στις λιγότερο αναπτυγμένες και τις πιο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πετύχαμε δηλαδή αυτή τη σύγκληση την οποία τη βρίσκουμε και μέσα σε μια ίδια χώρα χάρη στην κοινωνική προστασία. Αυτή η σύντομη περίοδος τώρα που έχουμε, από τότε που ξέσπασε η κρίση, έκανε το κοινωνικό μοντέλο να λειτουργήσει ανάποδα. Ε, λοιπόν, πρέπει αυτή η σύντομη περίοδος να μην επαναληφθεί. Και νομίζω ότι η μεγάλη δύναμη της Ευρώπης, ακόμα και οικονομικά μιλώντας, ήταν ακριβώς η δυνατότητά της να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και να φροντίσει όλες τις χώρε να αναπτυχθούν και να φτάσουν στα πιο ψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Σε αυτή τη λογική την οικονομική πρέπει να συνεχίσουμε να πορευόμαστε και θα το πετύχουμε αν βάλουμε την κοινωνική διάσταση στο ίδιο επίπεδο με την οικονομική. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιμιέ. Όπως εμφωνήσαμε και στην αρχή, τώρα θα δώσω την Προεδρία στην κυρία Ουλσκόκ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φιλίπ Κοντερί από την Γαλλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ χάρηκα που άκουσα όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ τις δύο αυτές μέρες, αλλά νιώθω και τώρα που είπαμε ότι πρέπει να ανυψώσουμε την οικονομία μας μέσω επενδύσεων, Ξετάσαμε το θέμα της δημοσιονομικής αλληλεγγύης, την συνεργασία που όντως είναι αναγκαία. Πράγματι, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία για να έχουμε και πάλι οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά όμως θα είναι μάταια αν συνεχίζουμε να παραβλέπουμε δύο τομείς τους οποίους δεν υπάρχει συνεργασία και οι διαφορές είναι τεράστιες. Το ένα είναι η φορολογία, δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα, το ξέρω, και το άλλο είναι οι πολιτικές μισθών και εργασιακών συνθήκων. Από το 2012 ακούσαμε ο, πόσο σημαντική είναι η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε πρόκειται για εκείνες του Ιουλίου, είτε για το πιο πρόσφατο πρόγραμμα εργασίας της, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η κοινωνική διάσταση απουσιάζει η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης έκανε μία πρόταση με τρία σημεία που για μας είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, είναι το θέμα της κινητικότητας, της κοινωνικής προστασίας όταν μετακινείται ένας εργαζόμενος, ότι τα κοινωνικά δικαιώματα δηλαδή πρέπει να μεταφέρονται να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, αυτό το κοινωνικό dumping που τόσο πολύ ζημιώνει τους εργαζόμενους. Και αυτά, το είπε και ο Πιέρα Λαμουέ, πηγαίνουν χέρι-χέρι με έναν ελάχιστο μισθό που να υπάρχει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερο στοιχείο είναι η συνέχιση της εγγύησης για την ολέα. Αν θέλουμε να πετύχει η εγγύηση αυτή για την ολέα, πρέπει να αναθεωρήσουμε την συγχρηματοδότηση και την προχρηματοδότηση, γιατί οι χώρες που βρίσκονται σε πιο δύναμη θέση είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο την ε, εγγύηση αυτή, οπότε πού να βρουν τα χρήματα. Τρίτον, επιδόματα αναργίας. Ένα ευρωπαϊκό πυλώνα που να μα επιτρέπει να μεταφέρονται τα επιδόματα αυτά από μια χώρα σε άλλη από εκείνη δηλαδή που έχει μεγαλύτερη άνεση προς μία που δυσκολεύεται περισσότερο. Ένα ευρωπαϊκό επίδομα ανεργίας θα βελτίωνε την οικονομική αποτελεσματικότητα της Ευρωζώνης, αλλά θα έδινε και νέα όθηση στην κοινωνική Ευρώπη. Θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους, αν προχωρούσε αυτή την ε, ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της πεντετούς της θητείας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σιμαντσίλια από την Λετωνία παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η οικονομική και φορολογική η πολιτική συνδέεται πολύ με τα κοινωνικά. Για τη Λετωνία η νομισματική ένωση αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών μας. Οι ανισότητες ανάπτυξης μεταξύ των χωρών, μελών και περιφερειών οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου ο πληθυσμός, όπου μειώνεται ο πληθυσμός στην Ήπεθρο. Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων είναι ένας μόνο τρόπος αντιμετώπισης είναι σημαντικό και ουσιώδες να να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία, η παράνομη εργασία. Επίσης και οι θέσεις εργασίας είναι σημαντικές αλλά και η ποιότητά τους, ιδιαίτερα επί τη βάση της επενδυτικής δέσμης. Και Πρέπει να τα συνδέσουμε όλα αυτά και με τις πιο ευάλωτες ομάδες. Γιατί υπάρχουν η ανισότητα των μισθών αλλά και η ανέχεια. Στην οικονομική πολιτική πρέπει να στοχεύουμε σε περισσότερη απασχόληση και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Να λεφτούν υπόψη και οι κοινωνικοί εταίροι και εθνικός και ενωσιακός. Ο κοινωνικός διάλογος είναι μέσον για να καταλήξουμε σε ανάπτυξη αλλά και στόχος καθεαυτόν. Γιατί έτσι αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι είναι τμήμα της κοινωνίας. Επίσης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν μεγάλη, μεγάλη δυνατότητα πρόοδου η Τσεχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε η Μαρίκα Όπστο για την κοινωνική διάσταση της κρίσης. Η ανταγωνιστικότητα στην ουσία φαίνεται μέσα από την μονιμότητα των θέσεων απασχόλησης. Εδώ και η καινοτομία και η παραγωγικότητα φυσικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης και υπάρχει και άλλη μία πλευρά η οποία δεν συζητιέται πάρα πολύ συχνά και η οποία αφορά στην ομοθεσία και στους κανόνες οι οποίοι πολλές φορές κάνουν τη ζωή δύσκολη στους επιχειρηματίες και στους παραγωγούς σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούμε εμείς να μειώνουμε συστηματικά τους μισθούς για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Παρ' όλα αυτά το κάναμε αυτό και επιτρέπουμε να γίνονται εξαγωγές προϊόντων από χώρες, εισαγωγές μάλλον, συγγνώμη, προϊόντων από χώρες οι οποίες παράγονται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Και ιδιαίτερα είναι κάτι που λειτουργεί υπέρ των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που αποφεύγουν να πληρώνουν το κοινωνικό κόστος της παραγωγής των προϊόντων τους. Έχουμε δύο επιλογές για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πρώτον, απαιτείται να εξετάσουμε προσεκτικά τους νόμους τους οποίους έχουμε περάσει σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε με χώρες οι οποίες παράγουν με ε, κοινωνικές αδυναμίες θα έλεγα. Πορτογάλος συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ποιότητα των παρουσιάσεων. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης είναι κάτι το πάρα πολύ αναγκαίο. Τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη μεταφράζονται κυρίως σε προβλήματα στον κοινωνικό τομέα. Απαιτείται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, και το ευρώ στην Πορτογαλία έχει μια ονομαστική αξία η οποία δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγική μας βάση και αυτό επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια κρίση η οποία επηρέασε την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Τώρα βλέπουμε ε, επιπτώσεις στον τομέα της υγείας, εξαιρετικά, μια εξαιρετική χειροτέρευση στις συνθήκες ζωής, εργασίας, διατροφής, παροχής υπηρεσιών υγείας, προβλήματα στον τομέα της πρόληψης, στον τομέα της υγείας, προβλήματα σε επίπεδο ψυχολογικό. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει τώρα να ακληθούμε, να διορθώσουμε. Ταυτόχρονα το ποσοστό των γεννήσεων ε, έχει αρχίσει να ε, μικρώνεται και προβλήματα δημιουργούνται ε, με περισσότερη οξύτητα στις περιφερειακές ζώνες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα διαφθορτικά ταμεία έτσι ώστε στον κοινωνικό τομέα τουλάχιστον να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο το ευρωπαϊκό πρότυπο να βοηθήσουμε τους νέους, να βοηθήσουμε τους ε, πολλού φτωχούς, ακριβώς όπως ε, το έχουμε κάνει ε, και με το Ταμείο της Συνοχής. Έτσι μόνο θα πετύχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση από τον Λόρδο Χάρισον, εργατικός από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω μαζί σας και με τον Λιθουανό συνάδελφο ότι η κοινωνική διάσταση θα έπρεπε να συζητηθεί ενωρίτερα. Θα ήθελα παρακαλώ να με διαβεβαιώσετε εσείς και οι συμπροεδροί σας ότι στην επόμενη διάσκεψη θα θέσετε το θέμα αυτό ενωρίτερα στην ημερήσια διάσταση. Ο Γκάι Ράιντερς μας εξήγησε γιατί πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και είπε ότι αντί να μιλάμε για τα stress test της κρίσης, μιλάμε για τα αντίστοιχα τέτοια τέστα για τις τράπεζες. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών είναι το πώς συνδυάζεται την κοινωνική διάσταση με τις οικονομικές ανησυχίες τις οποίες αναφερθήκατε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια πρακτικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Θέλω επίσης να συγχαρώ τη χώρα του κυρίου Ντομπρόφσκι, τη Λετωνία, η οποία πέρασε από τεράστια προβλήματα και πόνο για να μπορέσει να καταστήσει την οικονομία της πιο επιτυχή. Πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσετε κύριε Ντομπρόφσκι στην εμπειρία της χώρας σας. Ε, συνεννοείται και συμφωνεί για τα θέματα αυτά με τους κυρίους κυρίους Μοσχοβησί και Λόρτ Χίλ, τους συναδέλφους τους στην Επιτροπή. Η δική μου Επιτροπή και η Κάτω θέλουν να υπογραμμιστεί ακόμα μία φορά η κοινωνική διάσταση της λιτότητας οργανώνοντας ένα σεμινάριο για την λιτότητα. Θα σας αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες και έτσι πιστεύουμε ότι θα πάρουμε παραδείγματα από χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες ε, χώρες ε, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν την οικονομία τους να λειτουργήσει ε, ξανά. Μπορούμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτά, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα πάρετε τις απαντήσεις σας σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω όμως με τον κύριο Μιέ. Πιστεύετε ότι μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις κύριε Μιέ. Με μεγάλη χαρά. Αυτά έχουν απαντηθεί από την ιστορία. Πολλές φορές οι Ηνωμένε Πολιτείες του 1933 βγήκαν από την κρίση μέσω μιας κοινωνικής πολιτικής, το New Deal. Έβαλαν δηλαδή την κοινωνική προστασία μπροστά σε μια χώρα που δεν είχε καθόλου μέχρι τότε. Έβαλαν την πολιτική της απασχόλησης μπροστά σε μια χώρα που δεν την είχε καθόλου και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, από την αρχή δηλαδή της Ένωσης, όλοι μας πήραμε στοιχεία από το New Deal και τα βάλαμε στην πολιτική μας και έτσι δημιουργήθηκε η εποχή ανάπτυξης των 30 ετών από τον πόλεμο και μετά που τελείωσε με τον Bretton Woods που άρχισε με τον Μπρέντον Κούτς και που τελείωσε με την καταστροφή του. Και η ίδια είναι, πρέπει να είναι και τώρα η απάντηση. Αν μπορούμε να βάλουμε περισσότερη αλληλεγγύη μπροστά. Αν μπορούμε να βάλουμε τη σύγκληση μπροστά. Όπως είχε κατορθώσει να το κάνει μέχρι τώρα η Ευρώπη, τότε μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να συνδυάσουμε την οικονομία με τα κοινωνικά. Αν θέλουμε να πετύχει αυτό το πάντρεμα θυμάμαι μία φράση του Ζακ Ντελόρ που έλεγε αυτά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη είναι να συνδυάσει τον ανταγωνισμό και την μεγάλη αγορά με την αλληλεγγύη. Να οθεί και το άλλο ενισχύει. Αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή η δύναμη μιας οικονομίας είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο και πρέπει η Ευρώπη να μάθει ξανά να τα συνδυάζει αυτά τα δύο. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε Ντομπρόσκη, για πέστε μας σε τι ερωτήσεις θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλά σημαντικά ερωτήματα τέθηκαν πάλι και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα. Πολλά τέθηκαν για την κινητικότητα της εργασίας των εργαζομένων και από διάφορες απόψεις, από την άποψη του dumping, από την άποψη των μαζικών μεταναστευτικών ροών και της διαρροής ή ροής εγκεφάλων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Φέτος λοιπόν η Κομισιόν θα παρουσιάσει ε, μια δέσμη προτάσεων για την κινητικότητα των εργαζομένων. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή και να προωθήσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ροής ή διαρροής εγκεφάλων. Με καλύτερο συντονισμό των συστημάτων μας. Και αυτό σημαίνει και στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την κινητικότητα των εργαζομένων και μετά μερικά από τα ερωτήματα ξέφευγαν κάπως από το εύρος των υπάρχουσών προτάσεων όπως η κοινωνική διάσταση της νομισματικής ένωσης ας πούμε η ευρωπαϊκή ή ευρωπεριφέρεια ανεργίας και γι' αυτό έχουν συζητηθεί πολλές πρωτοβουλίες αλλά μερικές από αυτές uh, αλλά το κατά πόσον θα συμφωνηθούν αυτά εξαρτάται γιατί μπορεί να χρειάζεται αλλαγή των συνθήκων. Η Κομισιόν το εξετάζει αυτή τη στιγμή αυτό, αλλά μέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας συνθήκης, της ισχύουσας συνθήκης. Και θα δούμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε φυσικά. Πρέπει να υπάρξει και μία συζήτηση περισσότερο από τη στρατηγική σκοπιά, που και αυτή μπορεί να απαιτήσει αλλαγή των συνθήκων. Και φαντάζομαι ότι η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Αυτή η ευρωπαϊκή ασφάλιση για την ανεργία έχει συζητηθεί επίσης. Περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη συμμετοχή στους κινδύνους, ή mutualization όπως λένε όλο και περισσότερο, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει και περισσότερο έλεγχο, περισσότερο κόστος και περισσότερη παραχώρηση κυριαρχίας γιατί αν θέλουμε να αναλυφθεί περισσότερο να αναλυφθούν περισσότερο κοινή κίνδυνοι θα πρέπει να το αντισταθμίσουμε από κάπου αλλού. διότι όσο περισσότερο το συζητάμε τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι οι χώρες μέλη υπακούουν μεν στους ίδιους κανόνες αλλά εκχωρούν και περισσότερη κυριαρχία στην Ευρωπεριφέρεια. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με την ισχύουσα συνθήκη. Αυτό εξετάζουμε αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν. Και τώρα λίγο κάτι πιο προσωπικό για τους συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά τα έχω συζητήσει και με τον Επίτροπο Χίλ την εμπειρία μου στη Λετωνία, όχι μόνο. Αλλά δεν πρόκειται για ομοιόμορφες λύσεις για όλους. Πρέπει να δούμε και τα συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε χώρα και επίσης πρέπει να δούμε και τι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η προηγούμενη Κομισιόν, ας πούμε, είχε ασχοληθεί πολύ με θέματα οξέων οικονομικών και δημοσιονομικών κρίσεων και είχε βρει ορισμένες απαντήσεις, ενώ τώρα μιλάμε για τον κίνδυνο της πολύ αργής αναθέρμανσης, ανάκαμψης και τη δημιουργία <coughs> θέσεων εργασία. Αυτό που τελεί άλλες λύσεις διαφορετικές από τις προηγούμενες. Επομένως δεν είναι ομοιόμορφη λύση. Ευχαριστώ. Will Κυρία Μπάλτ, μήπως. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Στα πλαίσια της Προεδρίας μας η οργάνωση ε, τέτοιου είδους συναντήσεων την οργάνωση θα ακολουθήσει μια συνάντηση στις 23 Φεβρουαρίου στη Ρήγα. θα συμμετέχουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης των κρατών μελών και θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα της αγοράς εργασιας την κοινωνική ε, διάσταση της αγοράς εργασίας. Θα είναι παρόν ο Επίτροπος Ντομπρόφσκι, θα θέσει υπό την αιγίδα του τη συνάντηση αυτή Ελπίζω να δω όσους περισσότερους από εσά μπορώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ τη συνάντηση. Όσοι επιβιώσατε λοιπόν της διαδικασίας θαυμάζω το σθένο σας και λυπάμαι που το θέμα αυτό το κοινωνικό δεν το συζητήσαμε σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ και τον κύριο Ράιντερ. Σας ζητούν οι συμμετέχοντες να γίνεται η συζήτηση αυτή νωρίτερα στις επόμενες ε, συνεδριάσεις. Ελπίζω ότι και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πιο σοβαρά τώρα. Θα ήθελα να σχολιάσω. Αυτά που είπε ο Τσέχος συνάδελφος. Για κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν γίνεται εν κενό. Γίνεται σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Μιας παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας με διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες και εμπειρίες ανάκαμψης από την οικονομική κρίση. Και οι επιδόσεις οι δικές μας συγκρίνονται όχι με πολύ θετικό τρόπο για το, με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέξαμε εμείς στην Ευρώπη να αντιδράσουμε βασίζεται σε ορισμένες αξίες. Και μία από τις αξίες αυτές είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων γύρω από την απασχόληση. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 8. Αυτό δεν ισχύει για τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, κάτι πρέπει να λέει και για τις ε, διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά θέματα και η κοινωνική διάσταση των ε, εμπορικών συμφωνιών. Συνεπώς έχει σημασία ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ανταγωνιστικότητα με βάση τους χαμηλούς μισθούς και την απομείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και αναφέρομαι στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε με ικανοποιητικού ρυθμούς, με σωστά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και σε ένα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης σωστά και αυτοοργανωμένο. Και εδώ έρχεται το παράδοξο. Όλοι γνωρίζουμε τους κινδύνους που έχει ο τρόπος αυτός με τον οποίο επιδιώκουμε την ανταγωνιστικότητα. Ε, πρέπει να υπάρξουν διορθωτικά μέτρα όταν αυξάνεται ιδιαίτερο το κόστος παραγωγής, σαν παράδειγμα, και το κόστος εργασίας. Ξέρουμε το τι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Αλλά η αλλαγή αυτής της κατάστασης δεν είναι κάτι το εύκολο. Όταν μειώνεται το κόστος της εργασίας και μειώνεται το ποσοστό του κόστου στο τελικό προϊόν, δεν υπάρχει αυτόματη συλλογική διόρθωση σε σχέση με την οικονομική επίδοση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τελικά πολύ επικίνδυνο, πολύ πιο επικίνδυνο από την αύξηση των αμοιβών. Και μια και δεν γίνονται σε αυτό το επίπεδο διορθώσει, σε αυτό το τμήμα της εξίσωσης, αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα. Πώ θα ευθυγραμμιστεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και μέσω των μισθών είναι ε, το βασικό θέμα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε σε τομείς όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο καθορισμός των αμοιβών των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Έχω πάρει και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Δεν μπορώ να μπω τώρα πια σε λεπτομέρειες, αλλά εάν πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό, τότε θα πρέπει να επιδιώξουμε την καινοτομία και την αποδοτικότητα. Δεν μπορεί κανείς όμως να πετύχει αυτούς τους στόχους μέσω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας και μέσω της πληρωμής συστηματικά χαμηλών αμοιβών γιατί αν πληρώνει κανείς τους ανθρώπους σωστά για την εργασία τους, τότε θα πετύχει κανείς αποδοτικότητα και καινοτομία. Ο κύριος Ράιντερ το λέει καλύτερα από μένα αυτό, αλλά πάντως το θέμα της ανταγωνιστικότητας εδώ δεν είναι η μόνη λύση. Απαιτούνται σωστές συνθήκες εργασίας και σωστή αμοιβή. Τώρα για την νομοθεσία για το καμποτάζ. Νομίζω ότι καλή είναι η σκέψη, αλλά τα μέτρα που ελήφθησαν δεν λειτουργούν. Τώρα έχουμε ε, οδηγούς φορτηγών από τις Φιλιππίνες στις ευρωπαϊκές χώρες και στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Πληρώνονται ακόμα πιο χαμηλά και από αυτούς ε, τους οδηγούς από συγκεκριμένες χώρες μέλη. Δεν μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε ε, με τέτοιου είδους μέσα, την μείωση δηλαδή των αμοιβών και την μείωση των κοινωνικών συνθήκων. Γιατί τότε εμποδίζουμε την ανάπτυξη, εμποδίζουμε την αποδοτικότητα και θα διαλύσουμε ουσιαστικά την αίσθηση που θα θέλαμε να έχουν οι πολίτες στο εσωτερικό της Ένωσης. Ότι δηλαδή από κοινού θα δώσουμε τον αγώνα για σωστές συνθήκες εργασίας για τους πολίτες της Ένωσης. Έτσι θα οικοδομήσουμε την Ένωση. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ήσασταν όλοι αρκετά θαραλέοι που μείνατε μέχρι το τέλος αυτής της συζήτησης και όπως είπατε την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με την κοινωνική διάσταση. Δεν θα τερματίσουμε με αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ.